Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Uh, very warm welcome. Να σας καλωσορίσουμε θερμά μετά από τις ε, χριστουγεννιάτικες διακοπές. Αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Επομένως, καλή χρονιά σε όλους σας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω. Θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω ως συνήθως ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο μέσω web streaming και υπάρχει διερμηνία κατά προτεραιότητα στις γλώσσες των μελών της Επιτροπής μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση, θεωρώ ότι εγκρίνει τη μερίσια διάταξη. Και να περάσω τώρα στην έγκριση των πρακτικών. Έχετε στους φακέλους σας ε, τρία έγγραφα, πρακτικά της 12ης ε, Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, και της έκτακτης συνεδρίασης της 3ης Δεκεμβρίου. Μπορείτε να κάνετε παρατηρήσεις μέχρι το πέρας της σημερινής συνεδρίασης. Ε, εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρήσω ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Δεν υπάρχουν ε, κάποια άλλα σχόλια από πλευρά μου, επομένω επιτρέψτε μου να περάσω κατευθείαν στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Και επιτρέψτε μου να καλωσορίσω θερμά τον νέο πρόεδρο της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το στρατηγό Μιχαήλ Κωνσταράκο ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα το Νοέμβριο. αντικαθιστώντας ε, ένα στρατηγό ο οποίος είναι αρκετά γνωστός σε εμάς, ε, τον κύριο Ντερουσιέρ, ο οποίος συμμετείχε σε αρκετές συνεδριάσεις μας και είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε ε, συντομία το στρατηγό Κωνσταράκο τις πρώτες εβδομάδες ε, της θητείας του. Ήρθε και κατάφερε να επισκεφτεί και την πλειονότητα των ευρωπαϊκών αποστολών. Ε, συγχαρητήρια γι' αυτό. Στο σημείο αυτό το θέμα που μας απασχολεί είναι η στρατιωτική διάσταση της συνολικής προσέγγισης μια ανταλλαγή απόψεων με τον ε, στρατηγό τον κύριο Κωνσταράκο, πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατηγέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν ε, προχωρήσω στις παρατηρήσεις μου, θα ήθελα να σας ευχηθώ και σε εσά και στις οικογένειά σας ε, ό,τι καλύτερο για ένα ευτυχές ε, νέο έτος, επειδή είναι η πρώτη μας συνεδρίαση. Ελπίζω να ε, επιτύχετε σε όλες τις προσπάθειες. Είναι τιμή να έρχομαι εδώ σήμερα ενώπιάν σας, ε, ε, εφόσον είστε οι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης είναι τιμή μου να σας ενημερώσω για τις παρούσες στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Κυρίες και κύριοι, ο στρατός είναι ένα από τα αρκετά σημαντικά εργαλεία στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων. Ε, ένα αξιόπιστο και άμεσα διαθέσιμο εργαλείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές επιχειρήσεις ε, και αποστολές εν εξελίξη σε πολύ διαφορετικές ε, περιοχές και από γεωγραφική σκοπιάς. Γίνονται και στην Ήπειρό όπως γίνεται με την ε, ε, επιχείρηση EU4 Αλφία στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά και στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορά μας και τις γειτονικέ περιοχές, όπως για παράδειγμα ε, η επιχείρηση Uniformed Σοφία και η επιχείρηση Αταλάντη. Επίσης γίνονται και σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές τις οποίες αμφισβητούνται τα δικαιώματά μας και μπορεί η συνεισφορά μας να συνεισφέρει στο επίπεδο σταθερότητας, όπως για παράδειγμα στην αποστολή στο Μαλί και στη Σομαλία, ε, όπως επίσης και την επιχείρηση Αταλάντη, η οποία ε, είναι εξελίξη εκεί. Πάνω από 3.000 ε, στρατιωτικοί άνδρες και γυναίκες ε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή ε, σε διάφορες αποστολές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να διασφαλίσω στην Επιτροπή σας ότι αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα για μένα και φυσικά ε, ασχολούμαι πλήρω μαζί του. Γι' αυτό και ακριβώ επισκέφθηκα ήδη τι πέντε από τις έξι αποστολές ε, στο διάστημα των τριών μηνών περίπου από τότε που ανέλαβα καθήκοντα ω πρόεδρο τη Στρατιωτική Επιτροπή. Η έκτη είναι η επιχείρηση Αλφία στη Βοσνία Ερθεγοβίνη την οποία επισκέφθηκα πολλές φορές ε, κατά την άσκηση των προηγουμένων καθηκόντων μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω τώρα για κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, ξεκινώντας από τις ε, ε εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές. Αυτές οι αποστολές αποτελούν μια ανανέωση στη χρήση του στρατιωτικού εργαλείου και αυτό ε, είναι μια καινοτομία που θέλουμε να συνεχίσουμε και στο επόμενο διάστημα. Επιπλέον, η συνεισφορά του ε, στη συνολική προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική, όπω επίση και στη δημιουργία δυνατοτήτων στι ε, χώρε τις οποίε διεξάγονται οι αποστολέ μα. Η αποστολή στη Σομαλία ξεκίνησε το 2010 και παρά το γεγονό ότι αρχικά ε, ήμασταν στην Ουγγάντα, μετά όταν το επέτρεψαν οι συνθήκε, μεταφέρθηκε στο Μογκαντήσου γίνεται μια προσέγγιση τριών πυλώνων. Εκπαίδευση, συμβουλευτική διαδικασία και ε, βοήθεια, συνδρομή. Θέλουμε να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να έχουμε ειδική εκπαίδευση, ε, κυρίως μέσω μαθημάτων που γίνονται στο ε, στρατόπεδο εκπαίδευσης Τζαζίρα, κοντά στο Μογκαντήσου. Ε, μέχρι τώρα η UNAFOR Σομαλία έχει συνεισφέρει στην διάσωση, ε, στην εκπαίδευση 5.500 ε, Σομαλών στρατιωτών. Επίσης δίνονται συμβουλές στις Σομαλικές Αρχές ε, μέσω των υπηρεσιών ασφαλείας από το Υπουργείο άμυνα, δηλαδή και το Γενικό Στρατιωτικό Επιτελείο. Υπάρχει και το αρχηγείο στο ίδιο, στον ίδιο χώρο, υπάρχει μια αντιπροσωπεία εκεί και αυτό φυσικά θα μας δώσει τη δυνατότητα για αυξημένες συνέργειες και ενισχυμένη συνεργασία. Η αποστολή στο Μαλί ξεκίνησε το 2013, είναι αποστολή εκπαίδευσης, είναι επιτυχημένη και τώρα σε αυτή τη δεύτερη θητεία η οποία θα περατωθεί το Μάιο του 2016, οι 7 από τις 8 μονάδες μάχες ε, που προβλέπονται, οι GTIA στα γαλλικά, έχουν ήδη τύχη εκπαίδευσης. Ε, αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί... Ε, πιέζονται λόγω της ε, κατάστασης ε, ασφαλείας. Υπάρχει και η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, η ΜΙΣΜΑ, η οποία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο Συγγνώμη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία συμφωνίας και ε, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχουμε ίσως μία τρίτη θητεία για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αρχές του Μαλή αλλά να ε, ενισχύσουμε και όλη τη στρατιωτική ε, δυνατότητα της περιοχής. Μετά από την ολοκλήρωση της ε, ε, αποστολής EU4RCA το 2015 έχουμε πλέον μια συμβουλευτική αποστολή. Ο επικεφαλής της αποστολής έκανε πολύ σημαντική πρόοδο παρά τις πιέσεις που, που υπήρχαν και τους περιορισμούς. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με τη Μινούσκα την αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στρατηγική αναθεώρηση μαζί με τη διαδικασία διαχείρισης κρίσεων. Μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα στο ε, ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συγγνώμη, και εκεί ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια ακόμα επιτυχημένη ιστορία. Όπως γνωρίζετε, στις 7 Φεβρουαρίου θα γίνει ένας δεύτερος γύρος εκλογών και αυτή τη στιγμή θα υπάρχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, ε, θα είναι πολύ πιο εύκολη και η δική μας η δουλειά και θα μπορέσουμε ίσως ε, να αλλάξουμε την αποστολή μας ε, και να γίνει κάτι πιο απτό. Και τώρα να περάσουμε στις επιχειρήσεις. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη η επιχείρηση Αλθία δημιουργεί δυνατότητες και ταυτόχρονα παρέχει εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα ε, ενισχύει το περιβάλλον ασφάλειας ε, στη χώρα από το 2004. Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και αυτό φυσικά ε, σημαίνει ότι έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος και υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ της αποστολής και του αρχηγείου στο Σαράγεβο για να δημιουργήσουμε δυνατότητες και μονάδες μάχης στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιθωριοποιημένες ε, ομάδες ε, που αποτελούν ακόμα ε, παράγοντα στάθεια στη χώρα και πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Επομένως πρέπει να επαγρυπνούμε σε αυτή την περίπτωση. Η Ευρώπη ιστορικά εξαρτάται πάρα πολύ από τη θάλασσα. Το αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θαλάσσιος τομέας περιλαμβάνει ζωτικές πηγές της οικονομίας μας και φυσικά δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει και το γεγονός ότι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θαλάσσιες επιχειρήσεις. Στη Νότια Μεσόγειο έχουμε την αποστολή UNAFOR Σοφία από το περασμένο καλοκαίρι για να κάνουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες για να μπορέσουμε να ανακάψουμε την ε, ε, εμπορία ανθρώπων και να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο. Ε, αυτό είναι μόνο ε, μία διάσταση της προσπάθειας που γίνονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρώπινη τραγωδία που βλέπουμε να ξετυλίγεται στη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι και πολύ σημαντική συνεισφορά στην αποκατάσταση της σταθερότητας της περιοχής για η επιτυχία της αποστολής θα αυξήσει και τη δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών και των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο 2 της επιχείρησης, την ανοιχτή θάλασσα, που περιλαμβάνει ε, να, ε, το θέμα της αντιμετώπισης των σκαφών βάσει της απόφασης των ΗΕ του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του ε, ψηφίσματος 7 για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παράκτια κράτη, αν υπάρχει πρόσκληση των ε, λιβικών αρχών, να περάσουμε στη συνέχεια στο στάδιο 3. Τέλο, κατ' εξίσου σημαντικό, έχουμε την αποστολή Γιουναφόρα Ταλάντι, που ήταν η πρώτη θαλάσσια αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2008. Έκτοτε το επίπεδο τη πειρατεία ε, στι ακτές τη Ομαλία έχει μειωθεί ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πρέπει βέβαια να ε, καθησυχαστούμε. υπάρχουν και άλλες ε, προσπάθειες ε, για πειρατεία. Όλα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τη στιγμή που η διεθνή κοινότητα θα αποχωρήσει, οι ε, ναυτικές μονάδες που παρέχουν ασφάλεια στην περιοχή θα αποχωρήσουν, θα αναζωπηρωθεί η πειρατεία φυσικά και θεωρούμε ότι η αποστολή είχε πολύ μεγάλη επιτυχία για να μπορέσει να προστατεύσει τα σκάφη και να επιτρέπει την ασφαλή παράδοση πάνω από ένα ως εκατομμυρίου τόνων τροφίμων στις ακτές της Σομαλίας. Υπάρχουν ε, σχέσεις και με διάφορους διεθνούς παράγοντες όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Έθνη και τις διάφορες υπηρεσίες του, το ΝΑΤΟ, ε, τις ε, θαλάσσιες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες χώρες που ασχολούνται με την καταπολέμηση της πειρατείας. Είναι πολύ σημαντικέ επίση οι σχέσεις που ε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε με τον αυτιλιακό τομέα. Η UNAFOR Ατλάντα έχει συνεργαστεί και με το UCAP Nestor για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυνατότητε στην περιοχή και με άλλα ευρωπαϊκά όργανα και μέσα όπως για παράδειγμα το ε, πρόγραμμα θαλάσσιας ασφάλειας ε, μας. Θα πρέπει να γίνει μια ολιστική αναθεώρηση ε, της ε, ε, Αποστολής Ασφάλειας και Άμυνας ε, στη Σομαλία και στο κέρας της Αφρικής για να μπορέσουμε να δούμε τις δυνατότητες που είχαμε, τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε και πώς, τι έγινε με τις τρεις αποστολές στη Σομαλία ώστε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την περιοχή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό φυσικά μας δίνει και τη δυνατότητα να αποδείξουμε την αξία της ολιστικής προσέγγισης μας. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αποστολής έχουν και εννέα χώρες εταίρους εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Κάφκασος, ε, Γεωργία, Ευρώπη, Αλβανία, Φύρο, Μολδαβία, Ελβετία, ε, Τουρκία, ό, όλες αυτές οι χώρες συμβάλλουν ως προς το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Φαίνεται έτσι η βούλησή τους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες μας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Ενίσχυση των δεσμών με τον ΝΑΤΟ και με την, τον ΟΗΕ, με την Αφρικανική Ένωση, ε, συνεχίζεται, σημειώνεται πρόοδος, το ίδιο και ο διάλογος με τη ΣΥΠΑ, με την Αυστραλία, την Ινδία, το Πακιστάν, ε, τη Σερβία και ούτω καθεξής. Ε, ταυτόχρονα έχουμε διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με διάφορα μεμονωμένα κράτη, συνοριακά, Αλβανία, παραδείγματος χάρη, Φίωμ, Γεωργία κτλ οπότε βλέπουμε μια παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να είναι ελκυστικές οι αξίες μας. Δεν θα ήθελα να σας παραπλανήσω σε σχέση με τις επιχειρήσεις μας, να δώσω την εντύπωση ότι ε, λειτουργούν ε, χωρίς ε, προβλήματα και όλα βαίνουν αισίως. Ως συνήθως τα βασικότερα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε ως προς τη χρηματοδότηση Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ως προς ε, την εξασφάλιση των κονδυλίων ε, που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις εντοπισμένες ανάγκες. Στα πλαίσια της συνολικής ε, προσέγγισης έχουμε επίσης σημειώσει πρόοδο. Δεν πρόκειται για συγκεκριμένες ανάγκες διότι είναι μια προϊούσα διαδικασία. φυσικά υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στα πλαίσια της πρόληψης των συγκρούσεων και της ε, στρατιωτικής τεχνογνωσίας ε, θα πρέπει να αρχίζουμε τη δράση μας πολύ πρωτού ε, σημειωθεί, ξεσπάσει η κρίση και θα πρέπει να ξέρουμε ότι το στρατιωτικό εργαλείο είναι ευέλικτο, απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευράς ε, δυναμικότητας ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η συνολική στρατηγική για την, πολιτική, την εξωτερική πολιτική για την πολιτική ασφάλειας ε, θα, οι αποφάσει που λαμβάνουμε σήμερα θα επηρεάσουν κατά πολύ τις μελλοντικές μας δυνατότητες επίσης ένα συνολικό έγγραφο θα καλύψει όλες τις επιμερίες ε, στρατηγικές ε, και θα εξασφαλίσει και μεγαλύτερη συνοχή ε, ανάμεσα στις διάφορες δράσεις μας. Θα ήθελα για τις δυνατότητες που έχουμε να τονίσω τον σημαντικότατο ρόλο της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας σε βασικούς τομείς όπως τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, παραδείγματο χάρη επικοινωνίες με δορυφόρους, κυβερνοάμυνα και ούτω καθεξής, έχουμε χάρη σε αυτή την υπηρεσία ε, σημειώσει σημαντικότατη πρόοδο. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σημαντικό ο ρόλος της Στρατιωτικής Επιτροπής. ακόμη και αν αυτό γίνεται με ένα βελούδινο γάντι. Υπάρχει φυσικά η ήπια προσέγγιση η οποία συμπληρώνεται με τη στρατιωτική δράση και όπως σας είπα και νωρίτερα είναι ένα εργαλείο στρατιωτική δράση που είναι πάντοτε στην διάθεσή μας ε, και είναι ευέλικτο επίσης. Ε, μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ διαφορετικούς στόχους. Στόχους πολιτικές ε, ηγεσίας δεν είναι πανάκια για όλα τα προβλήματα, ούτε και πρέπει να είναι ίστατη λύση, διότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις για πολιτικά προβλήματα. Όμως, συγκεντρώνονται τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι πολιτικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να καταπολεμήσουν τις αιτίες της αστάθειας κατάρτιση, ε, συμβουλές προς τις αρχές σε κάθε χώρα είναι ένας βασικός ρόλος ε, ε, στο στρατιωτικό κομμάτι και Πιστεύω ότι αυτά ε, θα επιχούνται στην μελλοντική στρατηγική, συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί ε, σε λίγου μήνε. Ήδη έχουμε ε, στείλει τη συμβολή μα στην κατάρτιση αυτή τη νέα στρατηγική. Κλείνοντα, να πω ότι δεν είναι τυχαίο που έχουν ενωθεί οι ευρωπαϊκέ χώρε. Κάποιοι οραματιστέ πριν από κάποιε δεκαετίε θεώρησαν ότι δεν αξίζουν οι διαφορέ μα για να συνεχίσει ο πόλεμος στην Ευρώπη, όμως οι απειλές είναι ε, παντού και θα πρέπει να επιμένουμε σε αυτό που μας ενώνουν και σε αυτό που μας χωρίζουν. Αυτό είναι και η δύναμη της Ευρώπης. Η Ευρώπη υπάρχει επειδή υπάρχει πολιτική βούληση που εμπνέει τους πολίτες, τους οποίους εσείς εκπροσωπείτε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, σφαιρική αυτή παρουσίαση. Θα ήθελα τώρα να αρχίσει η συζήτηση. Ας ακούσουμε τον κύριο Αγνό Πρόεδρη, Πρόεδρε, στρατηγέ μου. Σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα τρει ερωτήσει να σα υποβάλω σε σχέση με συγκεκριμένε επιχειρήσει. Τα σχόλια είναι εκτό μικροφώνου. Ε, θα χρησιμοποιήσω τη συνεντεύξη σας για να βελτιώσω τα γαλλικά μου, αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, επιτρέψτε μου παρακαλώ να βάλω τα ακουστικά μου για να σας καταλάβω. Καλύτερα στα αγγλικά θέλω να ακούω, γιατί έτσι μπορώ να απαντήσω ευκολότερα. Δεν έχετε πρόβλημα πάντως. Ε, ε, πρέπει να μιλήσω γαλλικά, καταλάβετε μου για... γιατί θα με κατηγορήσουν μετά στην πατρίδα μου. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξή για κάτι που επανέρχεται συστηματικά στις συζητήσεις μας, το Ιράκ. Δεν μιλάω για τη Συρία, μιλάω για το, για το Ιράκ. Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες διμερώς παρεμβαίνουν είτε σε στρατιωτικές δράσεις, σε αεροπορικές επιθέσεις δηλαδή, είτε σε επιχειρήσεις αραγής ε, τεχνικής βοήθειας προς τον Ιρακινό στρατό και κυρίως βοηθώντας τους Πεσμέρκα, το κουρδικό κομμάτι και με προμήθειες εξοπλισμού. Αυτό αφορά ε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες και υποβάλλω το ερώτημα, ε, το τεχνικό κομμάτι του ερωτήματος αν θέλετε στο επίπεδο σας, ε, το επίπεδο της Στρατιωτικής Επιτροπής συζητείτε το ενδεχόμενο καλύτερο συντονισμού των επιμέρους μεμονωμένων δράσεων των κρατών στο Ιράκ. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια συντονισμένη δράση με συνέπεια σε σχέση με το, το στρατηγικό προσανατολισμό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, το άρθρο 42.7 της Συνθήκης Λισαμόνας θα επικαλέστε και πέρυσι πρώτη φορά η Γαλλία για την αμοιβαία αρρωγή, αμοιβαία αρρωγή ως προς την άμυνα των χωρών όταν δέχονται επίθεση. Ε, ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει η Στρατιωτική Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο. Και τρίτον, ένα διαρευνητικό ερώτημα. Διάφοροι Υπουργοί Εξωτερικών ή Υπουργοί Αμήνης ε, κρατών μελών, συγκεκριμένα ε, ισχυρών στρατιωτικά κρατών, Εσχάτως αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο ε, να γίνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη εάν ε, συγκεντρωθούν, όπως φαίνεται να συμβαίνει σήμερα, και οι πολιτικές προϋποθέσεις ε, με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερο για τον προγραμματισμό ενδεχόμενων τέτοιων επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Σκάν. Σας ευχαριστώ πολύ στρατηγέ για τα όσα είπατε. Κάποιες ερωτήσεις και θα ξεκινήσω και εγώ από την Λιβύη και τις ε, πρόσφατες εξελίξεις με την ε, κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης όσον αφορά την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, κάποια από τα προβλήματά τους, ε, ιδιαίτερα την αντιμετώπιση του ε, ISIS. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση σας και επίση. όσον αφορά την τρίτη φάση της επιχείρησης, πιστεύετε ότι θα δούμε πρόοδο και επίσης όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Βλέπουμε όλο και περισσότερες επιθέσεις οι οποίες επηρεάζουν τις κυβερνήσεις μας, ε, τις επιχειρήσεις μας και τους πολίτες ε, μας. Ε, τι σχέδια έχετε στον τομέα αυτών και τι γίνεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και επίσης υποθέτω ότι γνωρίζετε ότι θα υπάρξει δημοψήφισμα στο, στη Βρετανία. Ε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ανάλογα με το αποτέλεσμα και τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έχει στην άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το Αφγανιστάν. Είδαμε ότι η κατάσταση εκεί συνεχώς επιδεινώνεται, όλο και περισσότερες επιθέσεις από πλευράς των Ταλιμπάν. Ε, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις ε, στο Αφγανιστάν για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τζέφρι Βανόρτεν. Ευχαριστώ πολύ στρατηγέ. Συγχαρητήρια για την ανάληψη της θέσης αυτής. Αν και βέβαια είναι κάτι που έγινε ήδη πέρσι. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι σε τούτο το περιβάλλον ε, συχνά φανταζόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της αντιμετωπίζει τα ε, θέματα αυτά. Και ε, πιστεύουμε ότι αν δεν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνει τίποτα σε όλο τον κόσμο. Αλλά βέβαια αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Ένα από τους βασικούς τομεί ε, παρέμβαση τη ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι η Αφρική, όπου όμως επίσης ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε όπως και άλλοι κράτη ξεχωριστά, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κινητοποιήσουμε περισσότερο τους Αφρικανούς και ιδιαίτερα τις αφρικανικές ε, δυνάμεις ε, που έχουμε ε, σε εφεδρία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να ενισχύσουμε τις δυνάμεις αυτές και θα ήθελα να σας ρωτήσω και για ένα διαφορετικό θέμα. Πολλά λέγονται σχετικά με τον έλεγχο των συνόρων των χωρών μας, καθώς και τα νότια σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών. Στην στα παράλια της Μεσογείου. Τι οδηγίες έχετε λάβει εσείς όσον αφορά την εκπόνηση ε, σχεδίων επίγουσας ανάγκης για να ασφαλιστούν τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Μεσόγειο. Επίσης ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε στο ρόλο του EDA, του Οργανισμού Αμήνης. Υπάρχουν τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, ε, το θέμα της κυβερνοσφάλειας. Πολλά γίνονται από πλευράς των χωρών μας αλλά και από πλευράς του ΝΑΤΟ. Αλλά ε, το EDA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ε, πώς συμβάλλει σε όλα αυτά και πώς συμπληρώνουν αυτά τις εργασίες του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δάφμαν. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ στρατηγέ για την ε, ολοκληρωμένη παρουσίασή σας. Περιμένω... με ακούτε? Περι... Ωραία. Πάνω από 200 στρατιώτες από ό,τι κατάλαβα καλά ε, είναι τώρα συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρήσεις. πάνω από 3.000. Ε, ε, ξέρετε ότι ε, υπάρχει μια δημόσια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για την τρομοκρατία και ορισμένες φορές τονίζεται ιδιαίτερα το θέμα της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών. Ετίθεται το ζήτημα για τις υπηρεσίες πληροφοριών ε, στον στρατιωτικό τομέα. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε. Ο συνάδελφος επίση αναφέρθηκε πολύ σωστά στην πρόκληση που αντιμετωπίσουμε την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στο Στρασβούργο και αναρωτηθήκαμε ε, ε, ποιο θα είναι το μέλλον του Σέγγεν, Πώ θα εξασφαλιστεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων. Και εγώ αναρωτιέμαι, στο τομέα της άμυνας, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της. εμπόριο ανθρώπων διακινητές, ε, ποιος, ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούμε να αναλάβουμε, ποιες συστάσεις μπορείτε να εκπονήσετε, ώστε και σε αυτό το θέμα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων να μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική συμβολή. Τέλος. Αναφέρθηκαν ε, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη στον ενδεχόμενο ευρωπαϊκής ε, πολιτικής άμυνας και ποια είναι η ισχύς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε χρόνο και δεν χρειάζεται να σπέσουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα. Πιστεύετε ότι με ευρωπαϊκές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αναλυθούν ούτως ώστε η ευρωπαϊκή αμυντική κοινότητα να ε, ενισχυθεί. Τώρα, ε, είπε κάποιος συναδέλφος ε, για ότι επικαλέστηκε το άρθρο 47 η Γαλλία την περασμένη εβδομάδα. Συζητήσαμε με την είπατε εκπρόσωπο την κυρία Μογγερίνη και συζητήσαμε συγκεκριμένα για το ρόλο της Γαλλίας. Λέμε εκεί πως ε, ήταν πάρα πολύ θετικές οι αντιδράσεις όλων των κρατών μελών. Ε, η κυρία Μογκερίνη δεν θα μπορούσε η ίδια να επικαλεστεί αυτό το άρθρο ε, ζητώντας μια συγκεκριμένη επιχείρηση προωθώντας έτσι μια ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική στο μέλλον τι προβλέπετε ούτως ώστε να μπορέσει η ίδια η κυρία Μογκερίνη, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να επικαλείται αυτό το άρθρο και όχι ένα συγκεκριμένο κράτος όπως έγινε στην περίπτωση τη Γαλλία. Για την Αφρικανική Ένωση τώρα. Μας μιλάνε για μια δύναμη γενοκτονία στο Μπουρούντι. Επειδή είμαι Βελγίδα, ε, παρακολουθώ στενά αυτό το ζήτημα, έχοντας δει τι συνέβη στο παρελθόν στη Ρουάντα, θέλω να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε επί τόπου, τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε και ποια στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας ε, για αυτή την κρίση που απειλεί τη ζωή ε, του πληθυσμού του Μπουρούντι. Ε, στη συνέχεια θα σας στείλω και σχετικό mail. Ήθελα να ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ενδεχομένω να αντιμετωπίσει επιθέσει με χημικά και βιολογικά όπλα και πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την ετοιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Γκάλε. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε στην υποεπιτροπή μας. Θα ήθελα να μου κάνετε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το Μάλι και την αποστολή εκπαίδευσης που έχουμε εκεί. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου πείτε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πόσους έχουμε εκπαιδεύσει εκεί και πού έχουν ε, κινητοποιηθεί και επίσης πώς εξελίσσεται η συνεργασία στα βόρεια της χώρας ε, με τα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι κάποιες εκατοντάδες ε, Γερμανοί στρατιώτες επρόκειτο να σταλούν εκεί. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε τι στρατεύματα έχουν εκπαιδευτεί εκεί από εμάς. Και έχω μία ερώτηση για τη Βοσνία. Ε, η υποεπιτροπή επισκέφτηκε την χώρα πέρσι, μας εξήγησαν πώς έχει η κατάσταση. μα είπαν ότι έχουν περιοριστεί πολύ τα στρατεύματα εκεί και ότι σε τα χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται ασκήσεις. Υπάρχουν κάποια στρατεύματα εκτός Βοσνίας, αλλά ε, σε γειτονικέ περιοχές. Αναρωτιέμαι με βάση την πολιτική κατάσταση εκεί μήπως ε, θα έπρεπε να ενισχύσουμε τα στρατεύματα. Γνωρίζετε ότι η Σερβική Δημοκρατία, η Ρεπούμπλικα ε, Σερβσκα, έχει κάνει ε, κάποιες ε, είχε κάποιε δράσει εκεί πέρα και μήπω θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να προλάβουμε ε, ανεπιθύμητες ε, εκπλήξεις. Ε, και επίσης η Ελλάδα έχει σημαντικό στόλο και γνωρίζουμε ότι στα εξωτερικά σύνορα του Σέγγεν προς την Τουρκία πρέπει να διασφαλίσουμε τα σύνορα αυτά. Και επίσης, όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, μήπως θα ήταν δυνατόν η πολιτική να πει ότι θα διαθέσει μέρος ε, του στόλου για την προστασία των συνόρων και σε συνεργασία με την Frontex να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες του ελληνικού στόλου. διότι αλλιώς ε, τα σκάφη της Ελλάδας ε, απλά θα πλέουν ε, τη θάλασσα χωρίς όμως να διασφαλίζουν τα σύνορα. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ. Ε, στο τελευταίο, στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υπήρξε ένα ψήφισμα σε σχέση ε, με την ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 και στα πλαίσια αυτά υπήρχε και η, ο στόχος για τη δημιουργία μόνιμου πολιτικοστρατιωτικού αρχηγείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ενεργοποίησης του, του εν λόγω άρθρου ε, ποιος είναι ο ρόλος και η ε, αποστολή του συγκεκριμένου αρχηγείου ε, όπως τον επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ε, εκτιμάται ότι αυτό συνιστά, που εμείς το εκτιμούμε, ότι συνιστά επιθετικότητα, κλιμάκωση της επιθετικότητας και του χτυπήματος των λαών της περιοχής σε μια περίοδο που γενικά η όλη περιοχή μυρίζει μπαρούτι. Thank you. It was all from the floor. Ευχαριστώ. Ε, ολοκληρώσαμε με τις παρεμβάσεις. Θα ήθελα και εγώ να σας κάνω δύο ερωτήσεις, ε, στρατηγέ. Η μία είναι λίγο πιο γενική και αφορά την καταπολέμηση του ISIS, του Ισλαμικού κράτους. Δεν θα ήθελα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα ήθελα απλώς να μας πείτε ε, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς από κοινού ε, στην ενίσχυση της καταπολέμησης του Ισλαμικού κράτους, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι λίγο πιο συγκεκριμένη. Το περασμένο Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία ξεκίνησε. Έφτασαν στο Κίεβο. Θα πάνε στη Ταμπά, θα μείνουν εκεί για περίπου δύο εβδομάδες για να αξιολογήσουν την κατάσταση επιτόπου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, είπε στο διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην ε, ε, προηγούμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου ότι θα στείλει εκπρόσωπο στην Ουκρανία για να αξιολογήσει την κατάσταση. Υπάρχει και νέος επικεφαλής ε, της αποστολής στο Κιεβό, στην Πρόκειται για έναν εξαιρετικό Λιθουανό αστυνομικό. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει λίγο το πεδίο εφαρμογή και ο χαρακτήρας αυτής της αποστολή ή πρόκειται απλώ ε, για μια συνέχεια της κατάστασης που είχαμε μέχρι τώρα. Υπήρχαν ε, ζητήματα από την ε, Ουκρανία να αλλάξουμε και να διευρύνουμε λίγο το πεδίο εφαρμογής. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα ήθελα να είμαι λίγο σαφής. Το πιο σημαντικό εργαλείο, όπως σας είπα, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η συνολική προσέγγιση. Εγώ είμαι ένθερμος οπαδός της και αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει ό,τι παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση κρίσης ή ανάγκης. Και μπορεί ε, πολύ καλά να οριστεί με τον όρο Smart Power, ευφυής e δύναμη. Πρόκειται για ευφυή e δύναμη διότι είναι ένας συνδυασμός ε, ε ισχυρής και ήπιας δύναμης. Ε, η ισχυρή είναι το στρατιωτικό σκέλος και φυσικά οι ήπιες δυνάμεις είναι όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η συνολική προσέγγιση δεν είναι απλώς ε, άμυνα ή εκπαίδευση, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα ε, ανάπτυξη, κατάρτιση, το δικαστικό σκέλος, οτιδήποτε ε, μπορείτε να διανοηθείτε. Και αυτή είναι και η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ισχυρή ε, δύναμη ε, κατά τη χοντρική μου προσέγγιση είναι το πολύ 10%, μπορεί και λιγότερο. Ε, ίσως τώρα με τις νέες απειλές οι οποίες προέγυψαν ε, προέκυψαν προσφάτως μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο και μπορεί ίσως να χρειαστεί να φτάσουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό διότι οι απειλές είναι αναπάντεχες και δύσκολες ε, στην αντιμετώπιση τους. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και αν φτάσουμε σε ένα 20-25% είναι ήπια δύναμη, που σημαίνει ότι είναι όλα αυτά τα οποία ε, είναι πέραν του ελέγχου του δικού μου και ορισμένες φορές και των γνώσεών μου που σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να καλύψω όλες τις ερωτήσεις σας, ε, γιατί ε, εμπίπτουν σε αυτό το 85% των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς ε, δεν ε, είμαι σε θέση να πάω πέραν των πολιτικών μα ε, κατευθύνσεων. Δεν είμαι εδώ για να σας εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε είναι τι ακριβώς συμβαίνει στο στρατιωτικό τομέα. Όχι τι πιστεύει ένας στρατηγός για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός και αν δεν έχω αντιληφθεί σωστά το ρόλο μου. δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Θα ξεκινήσω λοιπόν ε, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις, μία προς μία, δραστηριότητες στο Ιράκ. Αυτές γίνονται σε διμερή βάση ή ε, σε ένα συνασπισμό αυτών που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν. Δεν έχουμε κάνει κάτι περισσότερο και δεν υπάρχει καμία συζήτηση, δεν έχω ακούσει τίποτα για ε, προσωπική μας εμπλοκή επιτόπου ή οποιαδήποτε δράση. Ε, εάν θέλετε να τα συνδυάσετε αυτά με το 42 ε, Παύλα 7, πρέπει να σας πω ότι η Γαλλία αποφάσισε διμερώς να ενεργοποιήσει το άρθρο και να έχει όλη τη βοήθεια που θα λάβει από τις διάφορες χώρες διμερώς. Είναι αλήθεια ότι ένας από τους τομείς ε, στους οποίους η Γαλλία ζήτησε συνδρομή ήταν η Συρία. Αλλά και αυτό ήταν σε διμερές επίπεδο. Επομένως, δεν έχουμε εμείς καμία αντίληψη της κατάστασης. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση για να δούμε πόσο επηρεάζει αυτό τις δικές μας τις αποστολές και τις επιχειρήσεις. Και επειδή στη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους ε, οι χώρες ε, μετακινούν ε, ε, στρατεύματα από το Μάλι στη Συρία είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και θα το συζητήσω με τις διάφορες χώρες. Αν οι διάφορες χώρες αποφασίσουν να ενισχύσουν τα θέματα για την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους χωρίς να επηρεάσουν τις δικές μας τις επιχειρήσεις ή ακόμα και τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών που είναι στην ίδια χώρα και παρέχουν ασφάλεια και σε εμά, τότε νομίζω ότι δεν είμαστε εμείς σε θέση να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Η είπατε εκπρόσωπος, η Φεντερίκα Μογκερίνη, νομίζω ότι εξήγησε πάρα πολύ καλά το ρόλο τον οποίο διαδραματίσαμε στο 42 ε, 7, καθώς επίσης και τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, ε, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση. Για τη Λιβύη. Για τη Λιβύη είμαστε στη φάση 2 που σημαίνει ότι έχουμε επιχειρήσει την ανοιχτή θάλασσα. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αποστολή μας θα πρέπει να πάμε ε, στη φάση 2 μπράβο που είναι επιχειρήσεις ε, στα λιβικά χωρικά ύδατα και στη φάση 3 που είναι ε, χερσαίες επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό, επειδή πάντα δρούμε με πάσα νομιμότητα, πρέπει να υπάρξει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και πρόσκληση από τις λιβικές αρχές. Και εκτός και αν μας δοθούν όλα αυτά δεν θα ξεκινήσει η επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι θεωρούμε ότι αυτά τα οποία κάνουμε τώρα δεν επαρκούν, απλώς διασώζουμε ε, ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πολύ σημαντικό. Σώζουμε ανθρώπινες ζωές και είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Αλλά αυτό ε, από επαγγελματικής και τεχνικής σκοπιάς δεν είναι αυτό που μας έχει ε, ζητηθεί να κάνουμε, που μας έχουν δοθεί εντολές οι λιβικέ αρχές ε, θα πρέπει να καταλήξουν σε γενική συμφωνία και η απόφαση ίσω να μας καλέσουν να δραστηριοποιηθούμε στα λιβικά χωρικά ύδατα και στη δική τους ε, την ε, ξηρά, εάν δεν υπάρξει δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε στη φάση 2 μπράβο και στη φάση 3. Για την κυβερνοάμυνα. Πράγματι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένας από τους τομείς στους οποίους ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσπαθεί να βελτιώσει τις δυνατότητές μας. Ε, είμαστε σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Ε, άλλωστε 22 από τα 28 κράτη-μέλη είναι κοινά μεταξύ των δύο διεθνών οργανισμών και συνεργάζονται λίγο πολύ, όχι σε όλα, αλλά σε πάρα πολλούς τομείς ε, στους οποίους ε, μας επιτρέπεται να συνεργαστούμε. Η κυβερνοάμυνα λοιπόν μας απασχολεί, συνεργαζόμαστε με τον ΝΑΤΟ και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ένας από τους τέσσερις τομείς των ευρωπαϊκών Δηματοτήτων στο, ε, και ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Όσον αφορά τώρα την πιθανότητα Brexit. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα επηρεάσει αυτό την, την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν μπορώ να σας πω και τι συνέπειες θα υπάρξουν. Διότι σε όλες τις επιχειρήσεις, ναι μεν υπάρχει συμμετοχή των ε, ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι σημαντικό σκέλος όλων των επιχειρήσεών μας, δεν κάνουμε όμως τέτοιες αξιολογήσεις. Ε, διότι ε, πρόκειται για κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί για τον οποιοδήποτε λόγο με οποιαδήποτε εκ των χωρών. Αν για παράδειγμα η Ελλάδα αποφασίσει να αποσυρθεί από μια επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο, θα προσπαθήσουμε ε, να κάνουμε μια διάσκεψη ε, για να αντικαταστήσουμε τις δυνατότητες οι οποίες αποχωρούν. Αυτό θα κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα με το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι η συνεισφορά των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρκετά ουσιαστική. Δεν ε, μας απασχολεί όμως αυτό το ενδεχόμενο προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Εξ όσων γνωρίζω, οι στρατιωτικές μας δυνάμεις δεν δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν, επομένως δεν μπορώ να σας πω τίποτα για το τι κάνουμε του Ταλιμπάν και δεν μπορώ να απαντήσω και ποιε είναι οι πολιτικές κινήσεις ε, εκεί τα, ε, πού συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο είναι το επίπεδο συμμετοχή. Νομίζω ότι έπρεπε να είχατε ρωτήσει την είπατε εκπρόσωπο την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε ε, στρατιωτικό ε, προσωπικό στο Αφγανιστάν. Τώρα, Αφρική. Ναι, εκεί έχουμε ιδιαίτερη συμμετοχή. Και γιατί έχουμε ιδιαίτερη συμμετοχή, διότι θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια και σταθερότητα στις χώρες ε, ε, στις οποίες έχουμε συμμετοχή και αυτό φυσικά απαντά και στην ερώτηση για το Μαλί. Διότι πέραν των πολιτικών προβλημάτων που έχουν και την πιθανότητα εμφυλίου πολέμου, γενοκτονίας και το καθεξής, ε, εδώ ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με άλλους οργανισμούς ώστε να μπορέσουμε να το αποφύγουμε, να το σταματήσουμε, να το ελέγξουμε. Επίσης όμως, ίσως αυτό το οποίο δεν γίνεται αντιληπτό εδώ, είναι ότι οι περισσότερες χώρες είναι δημογραφικές βόμβες, που σημαίνει ότι έχουν 6, 7, 8 ή και 9 παιδιά ανά οικογένεια, που σημαίνει ότι σε 10 χρόνια θα έχουν τριπλασιάσει τον πληθυσμό τους. Επειδή όμως δεν αναμένεται ταυτόχρονα να τριπλασιάσουν ή έστω να αυξήσουν τις δυνατότητές τους, τους πόρους τους, ε, θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Πρόκειται για χώρες με 80% αγράμματο πληθυσμό που έχουν μόνο ένα όπλο στα χέρια τους, αυτό το μόνο στοιχείο ενεργητικό που διαθέτουν. Είναι σαν οι δικοί μας οι νέοι να έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί έχουν όπλο. Αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα να τους προσλάβουν κάπου και να βγάλουν χρήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά δεν συνεισφέρουν σε καμία περίπτωση στη σταθερότητα επιτόπου και ε, στην ευρύτερη σταθερότητα της περιοχής. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον προκειμένου να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους, την ποιότητα ζωής τους, ε, την ίδια τη ζωή τους και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι ε, ξεκινούμε τους πολέμους, είμαστε σε εκπαιδευτικές αποστολές, εκπαιδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, για να έχουν ένα κατάλληλο στρατό, επαγγελματικό στρατό που ελέγχεται από δημοκρατικές κυβερνήσεις, στρατούς οι οποίοι δεν θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους ο βιασμός, στρατούς που δεν εκτελούν φυλακισμένους γιατί έτσι τους αρέσει ή γιατί είναι αστείο ε, και ευχάριστο αλλά ε, έτσι προσπαθούμε να επηρεάσουμε λίγο την νοοτροπία, ε, του στρατιωτική νοοτροπία στους τομείς αυτούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερο στο Μάλι ε, και τώρα θα επεκταθούμε και στις άλλες αποστολές, ε, θα το επεκτείνουμε και στο βαθμό που το έχουμε στο Μάλι, δηλαδή ε, να υπάρχει ανθρωπιστικό δίκαιο, να γίνονται μαθήματα ανθρωπιστική δικαίου και να γίνεται και σχετική εκπαίδευση να υπάρχει ένας κώδικας ε, διοντολογίας. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος να μου πει, ωραία, και τι νομίζεις ότι την επόμενη φορά που θα ε, ε, αρχίσουν να πολεμούν θα θυμηθούν όλα όσα τους είπες και θα σταματήσουν να θεωρούν προνόμιο τους κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ την ανθρώπινη φύση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από την εκπαίδευση αυτή θα γνωρίζουν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο καλό και στο κακό και θα ξέρουν ότι εάν καταστρέψουν ένα χωριό ή εάν ξεκινήσουν μια γενοκτονία μπορεί σε 2, 3, 4 χρόνια κάποιος οργανισμός, ευρωπαϊκός, ε, διεθνής, θα τους χτυπήσει την πόρτα και θα τους κατηγορήσει για εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν. Δεν θέλω να έχουν καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τελικά όταν βρεθούν στο πεδίο μάχη, ε, ούτε περιμένω να γίνουν θαύματα. Θέλω όμως να γνωρίζουν και αυτό σίγουρα θα επηρεάσει κάποιους από αυτού. Άλλωστε ε, βλέπουμε τρομακτικά περιστατικά και στην Ευρώπη, όπου ο κόσμος γνωρίζει ε, τι είναι έγκλημα και τι δεν είναι και παρόλα αυτά διαπράττουν εγκλήματα. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με μη κυβερνητικού οργανισμούς στον τομέα τον ανθρωπιστικό και θέλουμε να ε, διδάξουμε αυτή την οτροπία στους ανθρώπους, διότι πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Είναι κάτι που επηρεάζει, που επηρεάζει όχι μόνο τα στρατεύματα, αλλά και τον πληθυσμό γενικά. Και ο γενικός πληθυσμός είναι αθώος. Και δυστυχώς πρόκειται συχνά για τον πληθυσμό της δικής τους χώρας. Δεν παρέχουμε όμως ασφάλεια. Τι συμβαίνει λοιπόν σε όλες τις χώρες που έχουμε κινητοποιηθεί, είτε έχουμε αποστολές ε, του, των Ηνωμένων Εθνών ή υπάρχουν στρατεύματα της Αφρικανικής Ένωσης που στηρίζουμε εμείς οικονομικά στη Σομαλία πληρώνουμε τους μισθούς της Άμισομ των ε, στρατευμάτων ε, της Αφρικανικής Ένωσης ε, που καταπολεμούν την τροποκρατική οργάνωση Al-Shabaab. Και τα στρατεύματα αυτά προέρχονται από την ίδια την περιοχή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν πολεμούν μόνο για την χώρα στην οποία έχουν σταλεί, αλλά πολεμούν και για, για το δικό τους ε, συμφέρον, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από γειτονικέ χώρες. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν να έχουμε πρόσθετα μέτρα για τα πρόσθετα αφρικανικά στρατεύματα. Κάνουμε πολλά όμως για τα αφρικανικά στρατεύματα που πολεμούν εκεί επί τόπου. Όσον αφορά το θέμα των συνόρων, η μετανάστευση δεν είναι μέρος του στρατιωτικού τομέα των στρατιωτικών αρμοδιοτήτων. Δεν ε, είναι κάτι που αφορά την ε, υπηρεσία ε, εξωτερικών δράσεων, είναι, κάτι, είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν Ανακατευόμαστε λοιπόν στο θέμα αυτό. Ξέρω όμως ότι κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει τα σύνορά της. Και ακριβώς αυτό κάνουν. Δεν είδα ποτέ καμιά οδηγία, καμιά εντολή να πάμε σε κάποια χώρα και να ε, κάνουμε τη δουλειά της ε, συνοριοφυλακής. οι συνοριοφύλακες ε, δεν είναι όλοι οι ακτοφύλακες, είναι αυτές μονάδες ε, επιβολής του νόμου, δεν ε, υπάγονται στο Υπουργείο Άμυνας. Υπάγονται σε άλλους οργανισμούς, σε άλλες αρχές. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου. Όχι, σκέφτηκα ότι τα σκάφη θα μπορούσαν να διαβιβαστούν στην ακτοφυλακή η πρόεδρος διακόπτη. Σε λίγο θα έχουμε τον δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Πρόκειται για αρμοδιότητε ε, κυριάρχων κρατών. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει κάτι διαφορετικό, αυτό θα είναι μια πολιτική απόφαση. Εμεί κάνουμε αυτό που μα ζητούν. Αυτό συμβαίνει και με την επιχείρηση Σοφία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει την επιχείρηση αυτή. Ο προκάτοχός μου και το στρατιωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν την επιχείρηση αυτή σε χρόνο μηδέν και το έκαναν μάλιστα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να εκτελούμε τις εντολές που μας δίνονται. Ανταλλαγή πληροφοριών, ναι. Οι πληροφορίες επίση, οι μυστικέ πληροφορίε αποτελούν επίση αρμοδιότητα των ε, κρατών και γίνεται πολλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών και ακόμα και με χώρους ετε, χώρες εταίρους εκτός της περιοχής μας. Η ανταλλαγή πληροφοριών βελτιώνεται συνεχώς. Στην αρχή υπήρχαν σημαντικοί περιορισμοί διότι υπάρχει ένα παλιό Η πληροφορία είναι γνώση, η γνώση είναι εξουσία και δεν θέλουμε να μοιραστούμε την εξουσία μας με κανέναν. Αυτό όμως έχει αλλάξει τώρα. Πολλές χώρες ανταλλάσσουν πληροφορίες διότι συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις απειλές. Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας ανταλλάσσουν πληροφορίες. με χώρες και νομίζω ότι απάντησα όσον αφορά τα σύνορα των χωρών. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ναι, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε στενά, προσπαθούμε να λύνουμε όλα τα θέματα που υπήρχαν στο παρελθόν και να συνεργαζόμαστε όσο γίνεται πιο στενά. Αυτή... Αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα που μας έχουν αναθέσει οι χώρες μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον τομέα αυτόν. Χαίρομαι διότι βλέπω ότι πολλές χώρες αντιλαμβάνονται ότι μια αδύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σημαίνει και ε, ΝΑΤΟ χωρίς πολύ δύναμη. Ε, αν λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας, μάλλον οποιαδήποτε ενίσχυση θα επηρεάσει και τους δύο αυτούς οργανισμούς. Τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Καταρχάς, ε, για να ε, επικαλεστούμε ε, τις δυνατότητες αυτές θα χρειαστεί κάποιο περιστατικό. Και η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας προβλέπει ανεξάρτητες αντιδράσεις, δεν είναι σαν την ρήτρα αλληλεγγύης. που προβλέπει παρέμβαση της Επιτροπής ή κάποια κεντρική παρέμβαση. προβλέπεται παροχή βοήθειας σε κάποια χώρα που έχει κάποιο πρόβλημα και θα συμμετάσχουμε στο βαθμό που επιθυμεί η χώρα αυτή να συμμετάσχουμε. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Στο Μπουρούντι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μη στρατιωτική παρέμβαση. Μπορώ να σας πω ότι πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις. Αυτά έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, προφανώς τα ξέρετε ήδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και να βρει πολιτικές λύσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται πολιτική λύση και να μην ξεχνάμε ότι ε, η στρατιωτική λύση είναι πάντα η ίστατη λύση. Δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτήν. Όταν όλα τα άλλα μέσα αποτύχουν, όταν η κατάσταση ξεφύγει εκτός ελέγχου, τότε θα πρέπει να προσφύγουμε στο στρατό. Όσον αφορά την ε, άμυνα απέναντι σε βιολογικά και χημικά όπλα. Πράγματι, τα όπλα αυτά είναι μια από τις δασικές απειλές που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν χώρες με μεγάλες ε, τέτοιες ε, δυνατότητες επειδή πιστεύουν ότι υπάρχει σημαντική και άμεση απειλή, ενώ άλλες χώρες δεν είναι εξίσου καλά προετοιμασμένες. Όσον αφορά το Μάλι, μπορώ να σας πω ότι είναι σημαντική η επιχείρηση αυτή, η οποία θα επηρεάσει και τις πέντε χώρες της ζώνης Σαχέλ. προβλέπονται μεγάλα εκπαιδευτικά κέντρα για τους λόγους που ήδη σας ε, περιέγραψα. Το Μάλι είναι σημαντική χώρα της περιοχής και κάνουμε εξαιρετική δουλειά εκεί. Η Γερμανία δίνει μεγάλη σημασία στην περιοχή αυτή. Πρόκειται μάλλον για την ε, σημαντικότερη προσπάθεια της Γερμανίας ε, στην Αφρική και είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά που κάνει η Γερμανία. Εκπαιδεύει στρατεύματα, μεικτά, επιτόπου, τα οποία κινητοποιούνται εκτός της δικής μας περιοχής και κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί. Ακόμα και αυτό είναι ένα πολύ καλό μοτίβο, διότι με ρωτάτε πόσους εκπαιδεύσει. Δεν έχει σημασία. Η μεμονωμένη εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σπάνιο στον χώρο της άμυνας. Εκπαιδεύουμε στρατεύματα, δεν ε, εκπαιδεύουμε άτομα και προσπαθούμε να δούμε πού βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Κωνσταράκος. Εξετάζουμε λοιπόν να δούμε πού βρίσκονται οι ομάδες πολεμιστών και ποια είναι η σύνθεσή τους. Γίνεται λοιπόν εξαιρετική δουλειά και ξέρω ότι οι δυνάμεις εκεί και στην Ινούσμα και στην UTM Μάλι θα ενισχυθούν από χώρες που θέλουν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους. Όσον αφορά τη Βοσνία, δεν συμμερίζομαι τη θέση σας. Πραγματοποιούνται κάποιες ασκήσεις, υπάρχουν τοπικά στρατεύματα, υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Δεν συμμερίζομαι τη θέση σας όμως ότι θα βρεθούμε προεκπλήξεως εκεί. ή ότι θα έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε την δεκαετία του 90. Αυτή τη στιγμή δεν ε, βλέπουμε την ε, ανάγκη να έχουμε περισσότερους, ε, περισσότερες δυνάμεις εκεί. Όσον αφορά την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να μην πω τίποτα, διότι είναι η πατρίδα μας. Αλλά το θέμα των συνόρων είναι θέμα του κυρίαρχου κράτους. Είναι εθνική αρμοδιότητα. Όσον αφορά Ε, τα σύνορα και το μόνο που γνωρίζω είναι αυτό που γνωρίζω από τις ειδήσει. Ε, δεν έχετε κανέναν λόγο να φοβάστε. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα για ε, μόνιμη... για μόνιμο αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση του ΝΤΑΕΣ, Αυτή τη στιγμή έχουμε συμμαχία ε, εθελοντών, τη συμμαχία των πρόθυμων χωρών ε, και ε, στην Λιβύη δεν συμμετέχουμε λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στον αγώνα αυτόν και νομίζω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όπως σας είπα από την αρχή όμως, δεν συμμετέχουμε εμείς στην προσπάθεια αυτή. Ο στρατό επίσης δεν συμμετέχει σε καμία αποστολή στην Ουκρανία. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να σας πω τίποτα για το θέμα αυτό. Ε, δεν έχουμε τίποτα παραπάνω από τις έξι αποστολέ μας. Δεν ξέρω αν κάλυψα τις ερωτήσεις σας. Ξέρω ότι οι κύριοι Βανόρτεν και Γκάλερ θέλουν να κάνουν επερωτήσεις. Παρακαλώ. Μην ξεχνάτε ότι ε, λίγο ο γνώση που έχουμε στη διάθεσή μας για το επόμενο σημείο. Παρακαλώ να είστε συντομότεροι. Φανόρδεν, ευχαριστώ. Ε, συγκλονιστικά τα σχόλιά σας, ε, στρατηγέ. Νομίζω ότι απαντάτε με ειλικρίνεια. Ε, και δείχνεται τι γίνεται με αυτό το σύνδυο ε, με την πολιτική άμυνα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασόμαστε σε αυτή την εικονική έννοια, η οποία δεν ισχύει μόνο αποκλειστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και είναι και καινούργια ιδέα. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει, πολύ καιρό. Ε, είπατε μόνο το 10% αυτών των ε, περίεργων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στρατιωτικό σκέλος. Και είπατε ότι ουσιαστικά δεν ξέρετε τι συμβαίνει κατά τα λοιπά, διότι επικεντρώνεστε στο στρατιωτικό σκέλος. Ε, αυτό ε, τορπιλίζει την συνολική προσέγγιση. Ποια συνολική άμα δεν ξέρει η δεξιά, την πράτη, αριστερά και άλλο δεν ξέρουμε ποιος έχει ποιους πόρους. Αυτή είναι ε, η πραγματικότητα δυστυχώς. Για το άρθρο 42.7 και πάλι δείχνεται ότι είναι πολιτική μεθόδευση. Δεν είναι στρατιωτικός ο στόχος. Κανονικά η Γαλλία το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ έπρεπε να επικαλεστεί αν ε, το εννοούσε στα σοβαρά. Αλλά σωστά είπατε, ήθελε διμερή υποστήριξη και άρα έπρεπε να πάει από τα απευθεία στου άμεσα ενδιαφερόμενου και να τους πει θέλω βοήθεια επ' αυτού. Το 42-7 ήταν μια, ένα πολιτικό διάβημα, ξεκάθαρα. Για το Brexit δεν ε, το σχολιάζω, είναι, δεν είναι αμφίδρομη η διαδικασία, Αν δεν ήμασταν μέσα θα είχε φοβερό έλλειμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν επηρεάζονται οι ενοπλές δυνάμεις. Το αντίθετο μπορεί και να ε, επικεντρωθούμε και πάλι στην αναζωγόνηση του ΝΑΤΟ. Ε, μπορεί να μας βγει σε καλό αντί να καταστρέφουμε όλοι μαζί από κοινού αυτή την ε, αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αν ναι και να πω ότι στο Αφγανιστάν, ναι έχουμε Ιταλούς, Γερμανούς, Βρετανούς στρατιώτε. Ε, περίπου 500 έκαστος και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί ε, υποστήριξη, καν, κατάρτιση, καμία σχέση βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαίως. Το πλέον χρήσιμο στρατηγέ θα ήταν να την κλείσετε τη στρατιωτική επιτροπή και να ασχοληθούν όλοι με την αναζωγόνηση του ΝΑΤΟ. Αυτό χρειαζόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά για να χάνουμε το χρόνο μας. Okay, then I, I, I changed my questions Καλά, θα αλλάξω τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις μετά από αυτά που ακούσαμε. Ίσως συμφωνήσω το 42.7 είναι ε, πολιτικής εφήσης. Ε, το ίδιο όμως και το άρθρο 5. Ε, ποια είναι η διαφορά, είναι πιο ήπια η διατύπωση. Οπότε θα κερδίδαμε το άρθρο 5. Είναι πολιτική συζήτηση. Είναι ξεκάθαρο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πολιτική βούληση χρειάζεται και στι δύο περιπτώσει, αν κάποιος αποφασίσει να δράσει ή όχι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Χρηματοδοτικός μηχανισμός, ε, ο περίφημος ε, ή ο αποτρόπιος, πώς να το πω, μηχανισμός ε, Αθήνα για την χρηματοδότηση, νομίζω ότι αυτό συνιστά κόλλημα για την μεγαλύτερη συμμετοχή, διότι τι καλύπτονται, πάγια, 10%, που μπορούν να καλυφθούν από, αυτό το, αυτά τα μετρητά, το, το, ε, προς το κονδύλι που υπάρχει. Θα πιέσετε να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Βλέπω ότι κάνουν και δεν κάνουν τα κράτη-μέλη. Εσεί ε, όμω, επειδή έχετε τι τεχνικέ γνώσει και στην πράξη μπορείτε να κινηθείτε, δεν μπορείτε να μα πείτε πιο συγκεκριμένα ε, τι χρειάζεστε και να υποδείξετε από ποια κρατημέλη μπορείτε να το περιμένετε αυτό που χρειάζεστε. Δυστυχώ όμως ένα κράτος μέλος ε, πρέπει να καλύψει ε, όλα τα έξοδα παρότι ήταν ομόφωνη η απόφαση. Επειδή είστε ειδικό. θα ήθελα από σας να εξηγήσετε στους πολιτικούς ευθύνοντες τι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε αν ήταν ευρύτερη συμμετοχή και αν υπήρχε ένας επιμερισμός των δαπανών βάσει της κλίδας που έχουμε αποφασίσει. Πρόεδρος, ε, δυστυχώς πρέπει να κλείσει ο κατάλογος. Ξέρω, κυρία Ρότμαν, ότι πρέπει να θέλετε κι εσείς να συμμετάσχετε παρακαλώ μπορείτε να, να τα στείλετε γραπτός και να τα δει στη συνέχεια ο στρατηγός γιατί πρέπει να κλείσει τη συζήτηση ευχαριστώ για το δεύτερο γύρο. Για την ε, σφαιρική προσέγγιση. Σας είπα ότι ε, δεν προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες ασφαλείας, έχουμε τα τρία D ε, στα αγγλικά, ε, δηλαδή άμυνα, διπλωματία και ανάπτυξη νέων συστημάτων και μετά θα συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη του κράτους και στην ελπίδα που μπορεί να έχει για το μέλλον της. Δεν είμαι σίγουρος, όμως τελικά τι αποφάσισε η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει σε αφρικανικές χώρες, ποια κονδύλια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακή βοήθεια ή για οποιοδήποτε άλλο στόχο. Το ότι εγώ δεν έχω επίγνωση των κονδυλίων, όπως σας έλεγα προηγουμένως, ε, αυτό δεν σημαίνει πως υποβιβάζεται η αξία της ε, σφαιρικής προσέγγισης δεν ε, θυμάμαι σε χώρες, σε εθνικό επίπεδο, ο Υπουργός Αμήνης για να προσφέρει βοήθεια σε μια χώρα ε, παίρνει τηλέφωνο των διοικητή των ενόπλων δυνάμεων και τον, ε, τον ρωτά αν συμφωνεί. Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό σε κανένα κράτος. Εμάς μας ενημερώνουν όταν Πρέπει να προστατεύσουμε την επένδυση που έχει κάνει το κράτος. Δεν υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή και πρέπει να την ενισχύσουμε. Όχι αναπτύσσοντας εκεί νέες στρατιωτικές δυνάμεις, όχι βελτιώνοντας την κατάρτιση, τις δυνατότητες που έχουν οι δυνάμεις επιτόπου για να ε, κατοχυρωθεί η ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι χωλαίνει η σφαιρική προσέγγιση διότι δεν ενημερώνουν οι οργανισμοί που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ε, μονίμως τον ε, πρόεδρο της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής, όπως δεν σημαίνει και σε επίπεδο Υπουργού Αμήνης στα κράτη-μέλη. το άρθρο 42-7 σας απάντησα. Είναι ε, ήταν διμερής η ενέργεια, Μπορείτε να θεωρείτε ότι είναι πολιτικό διάβημα και να ε, τα συμπεράσματά σας. Μιλήσατε για το μηχανισμό Αθήνα. Αθηνά, συγγνώμη. Ε, για την ε, Πρόκειται για την κάλυψη δαπανών, ναι, αλλά ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος ο μηχανισμός με την πολιτική βούληση του κράτους. Ε, αυτό δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε, μπορούμε όμως να επηρεάσουμε το κόστος. Προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τους κανόνες ε, για την ε, χρηματοοικονομική εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις επιχειρήσεις, ε, όταν δηλαδή ζητούμε από χώρες να στείλουν στρατιώτες, είναι δύσκολο να το δεχτούν όταν δεν ε, προσφέρουμε κάποια οικονομική ε, ε, αποζημίωση να αντιστάθμισμα, διότι πολύ λίγες είναι αυτές οι χώρες που μπορούν ως εξαφνικά να διαθετήσουν εκεί τα μέσα τους επειδή κρίναμε εμείς ότι είναι σημαντικό, ε, σημαντική μια επιχείρηση και αρχίζουν να δαπανούν εκατομμύρια ξαφνικά επειδή το αποφασίσαμε εμείς. Υπάρχει όμως ε, έγκαιρα η προειδοποίηση και αυτό προσπαθούμε να επηρεάσουμε, δηλαδή να αλλάξουμε συνολικά το πλαίσιο του επιμερισμού ε, του οικονομικού άχθους. Αυτό το αντιγράψαμε από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, λέει, λέμε στο ΝΑΤΟ ότι ε, το κόστος σχετίζεται με, τον τομέα στον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια. Μπορεί κάποιος να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτός ο τομέας και άρα δεν θα πρόκειται να το χρηματοδοτήσω. Όχι, εμείς εντοπίζουμε τις ανάγκες ε, και τον εξοπλισμό ή τη δυναμικότητα που έχει κάθε κράτος μέλος και πώς μπορούν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν. Ε, αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η τη δυναμικοτητα που εχει καθε κρατος και πως μπορουν να καλυτερα να χρησιμοποιηθουν ε αυτο προσπαθουμε να αλλαξουμε ουτως ωστε να ειναι αποτελεσματικοτερη η συμμετοχη μας για τις ε, κοινοφελείς επιχειρήσεις ε, στις οποίες επιδόμαστε. Ευχαριστούμε. Ε, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Ευχόμαστε να μας ε, ξαναέρθετε σύντομα και να μοιραστούμε την εμπειρία που έχετε ε, στον τομέα αυτό. Κλείνει η συζήτηση και θα περάσουμε ε, ευθύ αμέσως στο επόμενο. Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Και να ξεκινήσω το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Και πριν σας ανακοινώσω τους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, ξέχασα να το πω αυτό, ε, στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Η κυρία Ελιζαμπέτα Πιέτο Μπόνο είναι πλέον επικεφαλής της Γραμματέας της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, ε, πρέπει να σας πω ότι ήταν εύκολη η μετάβαση και ελπίζουμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η κατάσταση στην ε, Ουκρανία, στην ε, EUEAM, την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε μαζί με την ε, ε, αντιπροσωπεία. Να καλωσορίσω την επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, της Ουκρανίας, την κυρία Πλέγκοβιτς και την, το διευθυντή Κένεθ Ντίν, ο οποίος μας είναι ιδιαίτερα οικείος. Ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, Διευθυντής της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων και την κυρία Λιούμπο ε, Νέποβ, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας καλωσορίσουμε σερμά Και να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Ντίν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρο, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας ενημερώσουμε σήμερα για την κατάσταση της πολιτικής αποστολής στην ε, Ουκρανία, την ε, ε, συμβουλευτική αποστολή. Ξέρετε ότι η αποστολή μας αποτελεί το ένα τμήμα των συνολικών προσπαθείς μας την Ουκρανία στον πολιτικό τομέα και γίνεται πολύ σωστά σε συνεργασία ε, και με άλλες οργανισμούς, ε, με άλλες αποστολές και υποστήριξη προς την Ουκρανία και φυσικά με τους διεθνείς εταίρους μας, ε, την USE, μια ειδική αποστολή παρακολούθησης και τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι λοιπόν τμήμα μιας ευρύτερης διεθνούς παρουσίας. Ε, δεν είναι έμνοπλη η αποστολή, για να σας επενθυμίσω, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 με πολύ συγκεκριμένο ε, δυνάμεις και υποστήριξη από την ε, Ουκρανία, από το Αρμόδιο Υπουργείο, ε, μαζί με τους Ουκρανούς εταίρους μας λοιπόν δραστηριοποιούμεθα. Ε, θέλουμε να έχουμε βιώσιμη ε, μεταρρύθμιση στην Ουκρανία, μεταρρύθμιση η οποία θα βοηθήσει στην επιβολή του νόμου με πιο αμερόληπτο, πιο νόμιμο τρόπο, ε, ώστε να μην υπάρχει απλώς εφαρμογή του νόμου και να υπάρχει πρόσβαση στους πολίτες στο νόμο, αλλά να βοηθήσουμε και την δημόσια εμπιστοσύνη ε, και φυσικά με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη πρόσφατα αναθεώρησαν την εντολή της αποστολής μας, την οποία θα σχολιάσω ε, εντός ολίγου αναλυτικά, αλλά με δύο λόγια η αναθεωρημένη αποστολή μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια στρατηγική εντολή η οποία θα συμπληρωθεί από πιο επιχειρησιακές στοιχές όσον αφορά την εφαρμογή του κράτους δικαίου επιτόπου. Αυτό εγκρίθηκε τον ε, περασμένο Ιανουάριο και η αποστολή θα έχει επιπλέον άλλα 140 άτομα, διεθνές προσωπικό και ε, τοπικό προσωπικό και επομένως ε, θα έχουμε μια αύξηση κατά 90 και κατά 7 άτομα αντίστοιχα, που είναι πολύ σημαντική ενίσχυση σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, τώρα υπάρχει ένας νέος επικεφαλής της αποστολής ε, στην ε, Βρυξέλλες. Ο νέος επικεφαλής θα αναλάβει καθήκοντα από Φεβρουαρίου ε, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σε σχέση με την αναθεωρημένη εντολή. Αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής της αστυνομίας ε, στο Βίλνιους ε, και αναπτύσσει προγράμματα στη Λεσουανία και η πυρογνωμοσύνη του κατά πάσα πιθανότητα θα βοηθήσει στην εφαρμογή αυτών που θέλουμε να κάνουμε. Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Φεβρουαρίου όπως σας είπα και ελπίζω ε, να μπορέσουμε να μιλήσουμε με όλους τους βασικούς μας συνομιλητούς τες από 1η έως 15 Φεβρουαρίου ώστε να ξεκινήσουμε σωστά. Είχα τη χαρά να ε, ε, συναντήσω και τον επικεφαλής αστυνομίας, τον κύριο Τεκνόητα, την περισμένη εβδομάδα. συζητήσαμε κάποιες εταιρικές, σκέψεις, εταιρικές σχέσεις από πλευράς μας. Θέλουμε να ε, βοηθήσουμε την ε, ειρηνευτική διαδικασία, σε καμία περίπτωση να την υποδαβλήσουμε και να προχωρήσουμε το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων ως εταίροι, ως αξιόπιστοι εταίροι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνομιλητές μας να προωθήσουν τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Το 2016 θα είναι κρίσιμη χρονιά για τις μεταρρυθμίσεις και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 2015. Να σας πω δύο λόγια για τις πέντε βασικές προτεραιότητες ε, για τη νέα επιχειρησιακή μας εστίαση αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταρχάς λοιπόν να έχουμε ε, καλύτερο ορισμό των αρμοδιοτήτων και των κανόνων και των ευθυνών ε, των βασικών θεσμικών οργάνων στην Ουκρανία. Το δεύτερο είναι η καλή αστυνόμηση, ε, αστυνόμηση της δημόσιας τάξης και ποινικέ διώξεις και εισαγγελικέ έρευνες και καθώς επίσης και τα ποινικά ζητήματα. Όλα αυτά θα συμπληρωθούν και από μια πιο μόνιμη παρουσία εκτός Κιέβου, ε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέχρι τώρα, αλλά δόθηκε ε, άδεια να υπάρχει παρουσία εκτός ε, της πρωτεύουσας ε, σε πιο στρατηγικό επίπεδο στα κρατη η αποστολή θα συμβουλεύει τις Ουκρανικές Αρχές σε ανώτατο επίπεδο ε, για το πώς θα μπορέσουν καλύτερα να τηρήσουν τους βασικούς κανόνες ε, για τα θέματα επιβολής του νόμου δεν θα πρέπει απλώς η κυβέρνηση να γνωρίζει τι συμβαίνει, αλλά να το γνωρίζουν και οι πολίτες. Και επομένως θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη λογοδοσία, μεγαλύτερη λογοδοσία της κυβέρνησης για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι αρχές επιβολής του νόμου όσον αφορά την αστυνόμευση, την προστασία των δικαιωμάτων, ε, παρακολούθηση και έλεγχο και θέματα εθνικής άμυνας, καθώς επίσης και τον ποινικό τομέα, το κράτος δικαίου και σε αυτά θα σταθώ εντό ολίγου. Είναι πολύ καλό λοιπόν να έχουμε τι σωστέ δομέ, τι σωστέ πολιτικέ και τι σωστέ στρατηγικέ ε, για να μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλη εποπτεία της διακυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο οι Ουκρανικές αρχές φροντίζουν να τηρείται το κράτος δικαίου για τους πολίτες τους. Ε, η αστυνόμευση μπορεί να ερμηνευτεί τώρα με διάφορους τρόπους, αλλά κυρίως ε, θέλουμε να συμπληρώσουμε αυτό που κάνουμε σε υψηλότερο επίπεδο, διότι η μεταρρύθμιση είναι καλή όταν οι πολίτες θα καταλάβουν τη διαφορετική, τη διαφορετική ε, νοοτροπία. Για παράδειγμα, το πώς τους μεταχειρίζονται οι αστυνομικοί ε, στα πλαίσια της νομιμότητας. Και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις με πιο απτό τρόπο ε, στη χώρα, σε όλη τη χώρα και να υπάρχει κατάλληλη ε, αστυνόμευση και να μπορούν να γνωρίζουν οι πολίτες τι υπηρεσίες μπορούν να τους παρέχουν ε, οι αστυνομικοί και σε τοπικό επίπεδο. Στο τρίτο στοιχείο τώρα, ε, δεν είναι τυχαίο το πώς επιλέγει, πρόκειται για διάφορους λόγους που οδήγησαν σε αυτόν, για παράδειγμα το Euromaidan και το πώς αντιμετώπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις στις ειρηνικές διαδηλώσεις. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς ε, να καταρτήσουν καλύτερα και να δώσουν καλύτερα εργαλεία για το πώς μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να κάνει μια ειρηνική διαδήλωση ε, χωρίς να καταλήξουμε σε περιστατικά βίας ε, στους δρόμους. Και πραγματικά θέλουμε να τους εκπαιδεύσουμε και να τους δείξουμε ε, πώς ε, μπορεί να χρησιμοποιείται αναλυγικά, νόμιμα και ε, κατά αύξονα βαθμό η ισχύς όταν χρειάζεται. Και φυσικά πρέπει να τους δώσουμε και τις δυνατότητες να το κάνουν, αλλά αναλογικά και στα πλαίσια του νόμου. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν καταλήλους αυτές τις καταστάσεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις διαδηλώσεις επιτόπου, αλλά να μιλήσουν και με τους διοργανωτές εκ των προτέρων για να μπορέσει να υπάρχει αμοιβαία συνεννόηση και από τις δύο πλευρές ε, για να υπάρχουν θέματα δικαιωμάτων και ευθυνών. Και αυτό είναι για να διασφαλίσουμε επίσης ότι κάθε φορά που διαπράτεται ένα έγκλημα μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στην αστυνομία για να καταγγείλει ένα γεγονός και η αστυνομία θα λάβει κατάλληλα μέτρα με σεβασμό των κανόνων, όπως τους κανόνες που ανέφερα στην αρχή ως πρώτη προτεραιότητα, για να υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και η πρόσβαση να καθορίζεται και βάσει αποδεικτικών στοιχείων, ε, και όχι με αυθαίρετες αξιολογήσεις ε, και με οικονομικά ε, ακατάλληλα κίνητρα. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα θέματα. Και τέλος υπάρχει και το θέμα της διαχείρισης των ανθρωπίνων ε, πόρων, ένα πιο ευαίσθητο θέμα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες ε, το κάνουν με ένωνομο τρόπο και με κατάλληλες δυνατότητες προαγωγής για τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και εργάζονται αμερόληπτα και νόμιμα. Ε, και να μπορέσει να υπάρχει πρόοδος και να μην υπάρχει νεποτισμός ή ε, κρατούμενο καθεστώς ε, επειδή ακριβώς κάποιος ε, είναι με τη σωστή πλευρά. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν κατάλληλη εκπαίδευση στο εσωτερικό επίπεδο, ώστε να επιβραβεύονται οι αστυνομικοί, αλλά να γίνεται και κατάλληλη διαχείριση και να μπορούν να παρέχουν κατάλληλα τις υπηρεσίες. Κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια ακόμα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος σε γενικές γραμμές θα ήθελα να πω ότι έχουμε κάποιε επιτυχημένες ιστορίες. Ε, μπορώ να δεχτώ φυσικά και επικρίσεις γιατί κάποια πράγματα δεν πήγαν όπως τα θέλαμε στην αποστολή του πρώτους μήνες. Αλλά η αποστολή ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη ε, σύνταξη του Εθνικού Νόμου για την Αστυνομία, γιατί αν δεν υπάρχει σωστός νόμος και σωστή στρατηγική, τότε δεν θα υπάρχει και κατάλληλη εφαρμογή και ε, δεν θέλουμε να γίνουν τα πράγματα λανθασμένα, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να κάνουμε τα σωστά πράγματα και να γίνουν σωστά όσα πρέπει να γίνουν και θέλουμε να είναι σωστός ο νόμος και να υπάρχει ισορροπία για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Ε, θέλουμε να έχουμε νέα αστυνομικά τμήματα, συμμετείχαμε πολύ σε αυτό για το πώς ε, θα λειτουργούν τα τμήματα αυτά. Ε, ε, μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε τα στατιστικά στοιχεία με διαφορετικό τρόπο, αλλά θέλουμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και το ευρύ κοινό να μπορεί να έχει καλύτερη πρόσβαση στην ε, τοπική αστυνομία. Ε, γίνεται αναθεώρηση επίσης του ποινικού κώδικα, τη στρατηγική για τα ε, νοριοφύλακες και θέλουμε να εξετάσουμε τις διάφορες πολιτικές. Και όλα αυτά γίνονται σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ, γιατί δεν θέλουμε να αναλάβουμε εμεί όλα τα καθήκοντα αυτά. Θεωρούμε ότι είμαστε ένα από του βασικού εταίρου, αλλά ένα από του πολλού βασικού εταίρου. Θέλουμε να διαδραματίσουμε επικοδομητικό ρόλο και δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα. Ε, πρέπει να κάνουν και οι εταίροι μα αυτά που του αναλογούν. Ολοκληρώνοντα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, η αποστολή θα διατηρήσει στρατηγικό ε, σχεδιασμό και θα επικεντρωθούμε στην καλύτερη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο με τα βασικά στοιχεία αυτά, ε, τα πέντε στοιχεία που σας ανέφερα και να υπάρχει κατάλληλη ε, κατανομή των ορμοδιοτήτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Νέποπ. Και θα ήθελα να ακούσουμε και τον κύριο Πλένκοβιτς. Εγώ παρετούμε από το χρόνο μου, δεν έχουμε εξαλλού ε, αρκετό χρόνο για τη συζήτηση. Νομίζω όμως ότι επειδή συμφωνούμε με τον κύριο Πλένκοβιτς ε, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Η κυρία Νέποπ, ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση της σημερινής ακρόασης στην Επιτροπή Αμήνης ε, και να ευχαριστήσω και την ε, Διακοινοβουλευτική ε, Επιτροπή. Είναι επίκαιρο το ζήτημα και είναι πολύ καλό που οργανώσατε τη σημερινή συνάντηση. Πολύ καλά τα είπατε κυρία Ντίν, καλύψατε ε, το ένα από τα κομμάτια που ήθελα να σχολιάσω και εγώ, οπότε μπορώ να επικεντρωθώ τώρα στο κομμάτι της ασφάλειας. Ε, συζητούμε λίγες ημέρες ε, μετά τις συζητήσεις που έγιναν για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, Γεωργίας και Μολδαβίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους υποστήριξαν το ψήφισμα μετά από τη συζήτηση. Νομίζω ξεκάθαρα φαίνεται μέσα από το ψήφισμα ότι ε, γίνεται αντιληπτή η κατάσταση στην Ουκρανία, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας ε, και απηχείται και το όραμα για τη μελλοντική μας δράση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξή της, την οποία εκτιμούμε δεόντως. Υπολογίζουμε εδώ και στη μελλοντική σας υποστήριξη και στην αλληλεγγύη και ενότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία είναι βασική προτεραιότητα για μας για να επιτύχουμε τον στόχο μας ως προς την ειρήνη και την αποκατάσταση εδαφικής ακεραιότητας ε, της χώρας μας ε, μαζί. Ευελπιστώ θα μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα εφέτος. Ε, και ε, ελπίζω να είναι θετικότερα το αποτελέσμα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Πέντε είναι τα σημεία ε, τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω εγώ στην ε, ομιλία μου. Για το γενικότερο πλαίσιο, για την κατάσταση επιτόπου στην Ουκρανία, θέλω να πω πως, όπως ακούσαμε και σε προηγούμενο τμήμα της συζήτησης για την σφαιρική νοηστική προσέγγιση, περί αυτού πρόκειται να μιλάμε για την ε, ασφάλεια. Και φυσικά για την Ουκρανία δεν μπορώ από το να αρχίσω με τον Τονβάς και την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ 2. Είναι ε, το πιο επώδυνο κομμάτι της συζήτηση και αυτό που κατεπηγόντως πρέπει να γίνει. Τελευταίες ημέρες ε, γίνονται θετικές δηλώσεις από τους εταίρους μας, όμως είναι πάρα ε, ευαίσθητη η θέση στην οποία βρισκόμαστε, συνεχίζονται οι επιθέσεις ε, και δεν μιλάμε καθόλου για την ε, κατάσταση στα σύνορα ε, ούτε για τα ρωσικά στρατεύματα, ούτε για τους ομήρους ε, και τους ε, κρατούμενους ε, που βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος. Δεν υπάρχει εκεί καμία πρόοδος και φυσικά ούτε και υπάρχει καμία πρόθεση να δοθεί ο έλεγχος των εδαφών της στην Ουκρανία. Ε, για την 20η Απριλίου δεν υπάρχει πρόθεση διεξαγωγής τοπικών εκλογών ανεξαρτήτως από την κατάσταση επιτόπου και θέλουν οι εκλογές να διεξαχθούν βάσει της ε, δική τους νομοθεσίας σε καμία περίπτωση δεν προτίθενται να ε, λάβουν υπόψη την, ουκρανική νομο, τον Ουκρανικό εκλογικό νόμο. Αυτό φυσικά συνιστά παραβίαση της σύμφωσης συμφωνίας του Μίνσκ είναι σε κρίσιμο σημείο η, διαδικασία. Δεν μπορώ να πω όμως ότι είμαι απελπισμένη. Δεν μπορεί να επιστραφεί το πάς. Αλλιώ δεν πρόκειται να λειτουργήσει η συμφωνία του Μίνσκ. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση ε, στους Ρώσους και όσους τους υποστηρίζουν για να εφαρμόσουν τη συμφωνία. Με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν πέρυσι πιστεύω ε, σημειώθηκε πρόοδος για την ε, διότι δόθηκαν αυτές αποδείξεις για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, τι μέλη γενέστε. Πρέπει να έχουμε ε, ξεκάθαρο χρονικό ορίζοντα για την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ, διότι ήταν προ... είχε προβλεφθεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του 2015, δεν έγινε αυτό. Πρέπει να ε, αποφύγουμε τις αλληλοκατηγορίες και τις χειραγωγήσεις, ε, τις ε, πολιτικές μεθοδεύσεις. Ε, νομίζω ότι η κατάβαση του πυρός ε, είναι το πρώτο που πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης, ο εκλογικός νόμος βάσει τον οποίο θα διεξαχθούν οι τοπικές εκλογές. Δεν περιμένουμε ε, την τελειότητα, δεν θα ήταν ρεαλιστικό, όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ουκρανίας πρέπει να συμμετάσχουν βάσει των προτύπων του ΩΣΑ και όπως προβλέπεται και από τη συμφωνία του Μίνσκ. Μετά, ε, όταν έχουμε τους αρετούς ε, προσωπούς, τι θα γίνει με ε, τα όργανα, με τις αρχές που υπάρχουν ήδη επί τόπου. Φυσικά, χρειαζόμαστε πολιτική υποστήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διεύρυνση της ε, ε, διεθνούς παρουσίας ε, επιτόπου. Ευχαριστούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμα την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με μια επιχείρηση ε, κοινής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας για την υποστήριξη της εφαρμογής των συμφωνιών του ΜΙΣΚ Πέρα από αυτό έχουμε και το θέμα της κατοχήρωσης του ελέγχου των συνόρων ε, αφού εφαρμοστούν οι συμφωνίες. Είμαστε ανοιχτοί, ε, συζητούμε επικοδομητικά και δείχνουμε ευελιξία στη σχέση μας με τα κράτη-μέλη και με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να, σε σχέση με την εντολή μιας τέτοιας αποστολής και την ε, ε, τα σχήματα βάσει των οποίων μπορεί να οργανωθεί. Θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο σημείο. Κρυμαία. Ε, πολιτική με αναγνώριση από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε και το εκτιμούμε. Τώρα πρέπει να δούμε πώ εφαρμόζονται στην πράξη αυτέ οι πολιτικέ. Ξέρετε ότι πρόσφατα ο πρόεδρός μας σκέφτηκε ε, να ψάχνει ε, τελικά αυτές τις λύσεις στο σχήμα Γενέβης 4 με την είπατε πρόσωπο να συμμετέχει ε, και η Ρωσία έχει δεχτεί, ε, ε, συγγνώμη, ασκείται βοηθή στη Ρωσία για να δεχτεί αυτή την πρωτοβουλία. με την παράνομη αυτή προσάρτηση ε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε φυσικά ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο της ασφάλειας και το, ε, που συνδέεται με την εδαφική μας ακεραιότητα. Δεν μπορούμε ε, να συνεχίσουμε όπως παλιά. Δεν μπορούμε όμως ε, ούτε και να διακόψουμε ε, τις διπλωματικές σχέσεις με την Ρωσία λόγω της εκκριμέας. Όμως θα πρέπει συνεχώς να το έχουμε κατά νου αυτό το σημείο. Τρίτο σημείο, μεταρρυθμίσεις. Μιλάμε για την επιχείρηση, η UAM, για την παρακολούθηση ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, πρέπει να είναι επικαιροποιημένη η εντολή αυτή τη επιχείρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας των πολιτών στην ε, Ουκρανία. Υπάρχουν ε, επίουσες ανάγκες για την ασφάλεια και χρειαζόμαστε αποτελέσματα με μια ενισχυμένη εντολή ελπίζω χάρη σε αυτή την επιχείρηση να μπορέσουμε να αναφέρουμε νέα πρόοδο. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό <clears throat> να ε, μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα ε, σχέδια για την ενίσχυση των πολιτικών αρχών. Τέταρτον, η οικονομική ασφάλεια. Έχουμε ήδη πολύ, καλές, ε, πολύ καλά αποτελέσματα. Ε, χάρη στην ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σίνκιβ θα παρουσιάσει συγκεκριμένες επιδόσεις, είναι ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας. Ελπίζω να μπορέσετε να παρευρεθείτε σε αυτή την εκδήλωση. Για τις μεταρρυθμίσεις θέλω να σας πω επίσης, σε σχέση με τη συμφωνία που κλείσαμε πέρσι με, την ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνης ε, ότι ανοίγει νέες δυνατότητες συνεργασίας ε, ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για την οικονομική ασφάλεια, κάτι άλλο εξίσου σημαντικό είναι η συμφωνία DCFTA. Ξέρετε πως το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας ανάμεσα στην Ένωση και την Ουκρανία είναι ότι η Ουκρανική οικονομία μπορεί να ακολουθήσει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και να λειτουργεί βάσει προτύπων που αποφασίζονται εδώ. Μπορούμε έτσι να εξυγχρονίσουμε την οικονομία μας. Τα περιοριστικά μέτρα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ε, λόγω της DCFTA συνιστούν ε, διακριτική μεταχείριση και είναι έκνομα. Ε, ο στόχος είναι να παρεμποδίσουν την Ουκρανία από το να εξυγχρονιστεί, να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Για να στεφτεί με επιτυχία η DCFTA Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα και ε, μην νομίζετε ότι θέλουμε να λειτουργήσει ως καθρέφτης, δηλαδή θέλουμε και εμείς ε, να κάνουμε αντίπινα κατά της Ρωσίας. Όχι. Θέλουμε να ε, είναι επιτυχημένες οι διμερείς μας ε, σχέσεις ε, και ε, ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Πέμπτο σημείο, απροφυγώς θα το σχολιάσω, ενεργειακή ασφάλεια. Ξέρετε ότι εφαρμόστε το πρώτο ενεργειακό πακέτο, χάρη στο οποίο μπορούν να έρθουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην, ευρωπαϊκή, ε, στην Ουκρανική ενεργειακή αγορά. Υπάρχει το θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου και της χρήσης ε, των ε, ε, δυνατοτήτων αποθήκευση που έχουν τα ταμιευτήρες μας. Υπάρχουν πολύ καλές δυνατότητες για την μεταφορά, τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου και για Ε, γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει να αποφύγουμε αγωγούς όπως ο Nord Stream που παρακάμπτουν την Ουκρανία. Πρέπει να εξυπηρετηθούν ε, οι ενεργειακοί στόχοι και από τις δύο πλευρές. Θα πρέπει να έχουμε μία πιο σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τους στόχους που έχουμε γενικότερα στις διμερείς μας σχέσεις. Κλείνοντας, ε, ε, υπολογίζουμε, θα έλεγα, στην ε, ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των συμφωνιών ΜΙΣΚΕ και την αποχώρηση της Ρωσίας από την Κρυμαία. Χρειαζόμαστε βοήθεια στις μεταρρυθμίσεις που κάνουμε ε, και ε, στην ε, πολιτική, οικονομική, ενεργειακή σφαίρα στον τομέα της άμυνας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα εργαλεία που έχουμε. Όπως είπε και ο στρατηγός Κωνσταράκος μιλώντας για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική, πρέπει να φέρουμε ασφάλεια και σταθερότητα και γι' αυτό εμπλεκόμαστε σε αυτή την περιοχή. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την Ουκρανία και άλλες γειτονικέ μας χώρες. Σας ευχαριστούμε και ξαναλέω υπολογίζουμε στη μελλοντική σας βοήθεια και παρουσία στην περιοχή. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Ανδρέη Πλένκοβιτς. επικεφαλή τη Αποστολή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φατίγα, ευχαριστώ κυρία Νέποπτε, κύριε Ντίν. Νομίζω ότι τονίσατε τα σημεία κλειδιά τη σημερινή συζήτησης που αφορούν όχι μόνο τη συμβουλευτική αποστολή αλλά ε, όλες τις πτυχές ασφαλείας της Ουκρανίας. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε συζήτηση για ε, το ψήφισμα για την σφαιρική και σε βάθος ζωνή ελεύθερων συναλλαγών. Νομίζω ότι ως θεσμικό όργανο καταφέραμε να αναλύσουμε επαρκώς την λεπτή θέση στην οποία βρίσκονται και οι τρεις χώρες και έχουμε και θα θέλαμε να εξανατονίσουμε την δέσμευσή μας για την δαφική σας ακαιρεότητα, αλλά να βοηθήσουμε και με αποστολές μας, ε, με ειρηνικό τρόπο την ε, επίλυση των ε, προβλημάτων. Όσον αφορά την ε, συμβουλευτική αποστολή, με μια σειρά αποστολών πέρσι και με την παρουσία πολλών συναδέλφων, είχαμε μια πολύ καλή επιτόπου ε, συνεργασία με τη Συμβουλευτική Αποστολή και με ε, τον ε, προηγούμενο επικεφαλής της Αποστολής. Από ό,τι κατάλαβα, ο κ. Λετσίνσκας θα ξεκινήσει τις εργασίες του αρχές Φεβρουαρίου. Γνωρίζουμε ότι είναι μια αποστολή η οποία μπορεί να δώσει περισσότερη ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα ασφαλείας είναι σαφής η επιθυμία να προχωρήσουμε πέρα από την εντολή που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή Ε, μέσω του, της αποστολής του ΟΣΕ να μην ε, περιοριστούμε σε συμβουλευτικό ρόλο, ο οποίος είναι φυσικά ε, πολύ χρήσιμος, αλλά να προχωρήσουμε και στην εποπτεία της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας, να παράσχουμε βοήθεια στην αστυνομία, στον δικαστικό τομέα. Νομίζω όμως ότι απαιτείται από εμά, δεδομένε και τι προηγούμενε ε, συζητήσει, ε, και για να αναφερθώ σε αυτά που ανέφεραν οι συνάδελφοι, ε, αναμένεται η κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας να είναι πιο παρούσα στην Ουκρανία. Μαζί λοιπόν με τις προτάσεις των χωρών υποδοχής και μαζί με την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκπόνηση εντολής της αποστολής που θα είναι κάτι ανάμεσα σε μια κλασική επιχείρηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, και ανάμεσα σε αυτό που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με την συμφωνία του Μίνς και υπήρξε συμφωνία του κουαρτέτου, του να παραταθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου η συμφωνία αυτή. Έτσι λοιπόν υπάρχει κίνητρο προς όλες τις πλευρές, για όλες τις πλευρές ε, να εργαστούν σκληρά για την επίτευξη των στόχων ε, της συμφωνίας. Υπάρχει λοιπόν έντονη διπλωματική ε, δραστηριότητα, επίσκεψη του Ρώσου εκπροσώπου στο Κίεβο και συναντήσεις ανάμεσα στην κυρία Νόλαντ και τον κύριο Σόρκοφ στην Ρωσία. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι υπάρχει επιθυμία να προχωρήσουμε για να βρούμε τρόπους ε, να εφαρμόσουμε τη συμφωνία του Μίνς, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, Ουκρανία. Ταυτόχρονα υπάρχει η συζήτηση για την ε, αποκέντρωση στο πλαίσιο της συνταγματικής διαπραγμάτευσης. Περιμένουμε τώρα τη δεύτερη ανάγνωση στην Ράτα και θα θέλαμε πολύ να δούμε η εφαρμογή της ε, συμφωνίας ε, του Μίνσκ ε, να συνοδεύεται από τα θέματα κλειδιά, δηλαδή η ειρήνη, δίκαιες εκλογές και με βάση την δήλωση που διάβασα σήμερα το πρωί δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ εύκολο να επιτευχθεί. Στόχος μας όμως είναι να σας βοηθήσουμε να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. Επίσης, ε, όσον αφορά την εφαρμογή της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, ε, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά και με την βοήθεια της ε, Επιτροπής μας για την ασφάλεια και την... τη βοήθεια της Επιτροπής μας της Ασφάλειας και Άμυνας θα μπορέσετε να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. Ε, να ανακοινώσω σήμερα, εκτός από την επίσκεψη του κυρίου Σίμκιφ αύριο, ότι θα διοργανωθεί τέλη Φεβρουαρίου, αρχέ Μαρτίου, εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 60 συνάδελφοι, 60 ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν ε, μεταξύ των οποίων ε, και οι επικεφαλής όλων των πολιτικών ομάδων και οι πρόεδροι όλων των επιτροπών για να δούμε πώς ε, μπορεί η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βοηθήσει στην οικοδόμηση ε, θεσμών στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ανδρέη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή των κοινών δραστηριοτήτων μας. Ε, κύριε Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. Θα μιλήσω γερμανικά, αν θέλετε φορέστε τα ακουστικά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τις ε, κοινέ αυτές δραστηριότητες ε, στην Ουκρανία και έτσι μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι κατά τον εξυγχρονισμό της χώρας και να ε, πραγματοποιήσουμε αυτά που περιμένει ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό να εξελιχθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα και ο κόσμος το νιώθει αυτό. ως Ευρωπαϊκή Ένωση με την αποστολή αυτή μπορούμε να επικεντρωθούμε σε θέματα που θα νιώσουν πολύ σύντομα οι πολίτες. Θα, πραγματοποιη... θα αλλάξει δηλαδή η πραγματικότητα για τους πολίτες επιτόπου, για παράδειγμα. Στην Τροχέα, στο Κίεβο και στην Οδυσσό. Είχαμε ε, εξυγχρονισμό του συστήματος ε, και έχει ε, φανεί ήδη αυτό το νέο πνεύμα της αστυνομίας. Επίσης, στην Οδυσσό έχουμε νέο πρόγραμμα. Τη δημιουργία ενός κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών. ώστε να μην είναι όπως παλιά που ε, έκλεινε κάποιος ραντεβού με έναν ε, υπάλληλο και ε, κλεινόταν σε ένα μικρό δωμάτιο που πιθανότατα να γινόταν και δωροδοκία. Τώρα λοιπόν αλλάζει το σύστημα και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί κανείς να κάνει τη δουλειά του. Συμμετέχουμε λοιπόν στην προσπάθεια ε, αλλαγής ε, της ζωής των ανθρώπων ε, και εξυγχρονισμού. Σε άλλους τομείς όμως όπως είναι η εσωτερική ασφάλεια, τι κάνουμε και τι κάνουμε όσον αφορά την τεχνική βοήθεια. Για παράδειγμα, πυροσβεστική. ή για άλλους οργανισμούς ε, για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ε, διότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα για τους ανθρώπους εκεί επί τόπου. Όσον αφορά τις εκλογές ε, στα κατεχόμενα εδάφη και την εφαρμογή της Συμφωνίας του και γενικά, γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι για τους φίλους μας από την Ουκρανία να είναι μάρτυρες ε, αλλαγής ε, του συντάγματος ε, στις περιοχές αυτές. Νομίζω όμως ότι από πολιτικής πλευράς είναι πολύ σημαντικό η Ουκρανία να εκπληρώσει το δικό της μέρος των υποχρεώσεων, ώστε κανείς εδώ στην Ευρώπη να μην μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση του τύπου ότι οι Ρώσοι ούτως ή άλλως δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και ούτε η Ουκρανοί. Έτσι λοιπόν μπορούμε να άρουμε τις κυρώσεις. Είναι σημαντικό η Ουκρανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την αλλαγή του συντάγματος. Άλλωστε πιστεύω ότι οι δυσκολίες είναι προσωρινές. Μόλις λήξει η κατοχή θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι άνθρωποι ε, σε μια φυσιολογική πραγματικότητα. Η πολιτική μου έκκληση όμως είναι από τη δική σας πλευρά να κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να μπορείτε να πείτε ότι τουλάχιστον η Συμφωνία Μίνσκ όσον αφορά τη δική μας ε, πλευρά έχει εφαρμοστεί. Ευχαριστώ κύριε Σφρόιντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για μένα τώρα, γιατί και ο κύριος Πλένκοβιτς και ο κύριος Γκάλερ ε, ουσιαστικά είπαν αυτά τα οποία ήθελα να πω και αυτά τα οποία ήθελα να επισημάνω. Θα είμαι λοιπόν πάρα πολύ σύντομο. Ε, συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα ακούστηκαν προηγουμένως. επομένω δεν θέλω να τα επαναλάβω όλα αυτά. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ είναι το πιο σημαντικό τμήμα ώστε να επιληθεί το ζήτημα. Και προχωρούν πολύ αργά, προχωρούν πολύ πιο αργά από ό,τι θα περιμέναμε, αλλά όπως γνωρίζουμε ε, πάντα υπάρχουν δύο μέρη σε μια ε, σύραξη, επομένως τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να συνεχίσω και από αυτά που είπαν ο κύριος Πλένκοβιτς και ο κύριος Γκάλερ και να σας ξαναρωτήσω μέχρι ποιου σημείου έχει προχωρήσει η Ουκρανία ώστε να αλλάξει την νομοθεσία περί ε, απόδοσης χάριτος που εξακολουθεί να αποτελεί ακαθόδε ζήτημα, τον εκλογικό νόμο και τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά βήματα τα οποία πρέπει να ε, κάνει η Ουκρανία και όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ, εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά επιθυμούμε να προχωρήσετε γρήγορα ε, στην επίλυση αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στιτίνα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κυρία Νέποπ, είπατε ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ είναι ο μόνος τρόπος για να επιληθεί το πρόβλημα ισχύει αυτό, διότι συζητούμε την κατοχή τμήματος της Ουκρανίας εδώ και δύο χρόνια και εδώ και δύο χρόνια πεθαίνουν άνθρωποι ε, και κοντά στο Ντούνιεξ και στο Σύριακ ε, υπάρχουν περίπου 1,5 ε, εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπισμένοι που δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Μέχρι ποιο σημείο λοιπόν θα ακούμε τις υποσχέσεις του κυρίου Πούτιν ε, ε, για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες άλλες λύσεις, άλλες οδοί. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Ποροσέγκο μας ζητά πολεμοφόδια ώστε να μπορέσουν να υπερασπιστούν τους αυτούς τους, ώστε να μπορέσουν να υπερασπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο ε, τις περιοχές τους. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσον ε, μπορείτε να θεωρείτε ότι και αυτές θα μπορούσαν να είναι λύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόνι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση η οποία σχετίζεται με το ουκρανικό ζήτημα, αλλά στέλνει και μηνύματα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις τελευταίες ε, δύο εβδομάδες Είδα ακόμα και σε τροπολογίες, ε, γραπτές προτάσεις, ε, το γεγονός ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός στο ρωσικό εμπάργο τροφίμων ε, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, αντάλλαγμα να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις. Ε, θα ήθελα εδώ να διορθώσω το εξής. οι κυρώσεις αφορούν την επίθεση στην Κρυμαία και δεν έχουν καμία σχέση με το εμπάργο των τροφίμων. Επομένως, ακόμα κι αν ε, κάποιος κάνει κατά λάθο μία ε, ανάμειξη των δύο καταστάσεων ε, θα δημιουργήσει προβλήματα και στο κοινοβούλιο. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ δράσεων ε, για να συνεχιστούν οι κυρώσεις όσο ε, θα τελεί υποκατεχεί η Κρυμαία από ρωσικά στρατεύματα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό με το εμπάργκο στα τρόφιμα. Ε, των Ρώσων ε, ε, από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ήθελα να το πω ως διευκρίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω και εγώ μια ερώτηση και στον Διευθυντή, τον κύριο Ντίν και στην κυρία Νέποπ. Καταρχάς, για τους ε, τρόπους ε, συνεργασίας ε, με την αποστολή του ΟΣΑ, πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε κύριε Κίν να ενισχύσουμε την παρουσία μας στα Ουκρανο-Ρωσικά σύνορα και τι δυνατότητες υπάρχουν. για να δράσουμε στην αποστολή αυτή, αν μπορεί η αποστολή UAM να ε, συνεισφέρει και αυτή από πλευρά της. Και προς την κυρία Νέποπ, από τις πρόσφατες εκθέσεις διαβάζουμε ότι υπάρχουν περίπου 8.500 ρωσικά στρατεύματα στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Τι προβλέπετε να γίνει. Είναι ένοπλοι ε, και έχετε και στρατεύματα εκεί. Τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια. Mr. Keane, please. I think that's it's all in terms of questions, so we can give the floor to, to both uh, Mr. Keane, the Director Keane and Madame Nepop. Στην Nepop και αν και ο Αντρέη θέλει το λόγο, παρακαλώ. Um, I, I, I might start with the... Θα αρχίσω με τα επιχειρησιακά ε, με το επιχειρησιακό κομμάτι και η συνάδελφος θα ασχοληθεί με το πολιτικό κομμάτι. Για την ειδική βοήθεια, κοιτάξτε, είναι βασικός ε, εταίρος ε, για την EUAM, όχι μόνο επειδή έχει τους άλλους βασικό ρόλο, αλλά διότι έχουμε το όργανο της ε, σταθερότητας και της ειρήνης ε, που πληρώνει τα δύο τρίτα της ε, χρηματοδότησης για αυτές τις επιχειρήσεις. Οπότε ε, σε μεγάλο βαθμό χάρη σε εκείνους μπορούμε να έχουμε αυτή την επιχειρηστές θωρακισμένα. Έχουμε 70 ε, οχήματα, έχουμε στο σύνολο 20 ε, από την Καμπούλ, γιατί είναι δύσκολη περιπολία στην ανατολική περιοχή. 30 οχήματα μη τεθωρακισμένα από το Κοσφοπέδιο και επίσης ε, έχουμε ε, ιατρικά κίτ, ε, διότι είναι πολύ δύσκολε οι αποστολέ στην περιοχή. Επίση, δορυφορικέ εικόνε για την, τον εντοπισμό των δυνάμεων για εξοπλισμό. Δηλαδή, είναι πολύ στενό εταίρο μα και για του πόρου, για τον εξοπλισμό, αλλά και για τα κονδύλια. Και έχουμε και ανθρώπου επιτόπου συγκεκριμένα που έρχονται από διάφορα κράτη-μέλη. Μία φορά την εβδομάδα σε επίπεδο τακτικής, αλλά και σε επίπεδο οργανώνονται και δεν υποστηρίζουν άμεσα τη Μίνσκα, αλλά πρέπει να ξέρουμε οι μεν τι κάνουν οι δε. Είναι στα πλαίσια της ε, διεθνούς προσπάθειάς μας ε, στην Ουκρανία και χρησιμοποιούμε τους πόρους ε, γιατί είναι σημαντική και είναι απαραίτητη για την περάτωση της δικής μας επιχείρησης για τις επιχειρήσεις προς τη φυσική καταστροφή, παραδείγματο χάρη και άλλου είδους επιχειρήσεις. Δεν είναι στα πλαίσια της εντολής μας, ε, διότι ασχολούμαστε με την πολιτική ασφάλεια και άμυνας και σε αυτό εντάσσεται η εντολή μας. Ε, αλλά ε, φυσικά θα πρέπει να προσφέρουμε συνολικές υπηρεσίες στο λαό της Ουκρανίας. Συμφωνώ μαζί σας. Σας είπα τα πέντε επιμέρους τμήματα ε, και για τον επιμερισμό των ευθυνών ε, ε, για την επιβολή του νόμου και τις αστυνομικές δυνάμεις υπάρχει η εντολή για τις στρατιωτικές δυνάμεις άλλη εντολή έχουν αυτοί άλλη εντολή έχουν οι αστυνομικές δυνάμεις Οπότε θα χρειάζεται καλύτερο ορισμός, ώστε να οριστούν ποιε είναι αυτέ οι αρχές επιβολή νόμου. Όταν μιλάμε για καθολικές υπηρεσίε ε, και στα πλαίσια μέσης εντολής ε, υπηρεσιών σε, κατάσταση επίγουσα ανάγκη. Έτσι μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Ένας καλύτερος ορισμός χρειάζεται λοιπόν και ως αποτέλεσμα θα προκύψουν καλύτερες υπηρεσίε. Για τη μεταρρύθμιση των αστυνομικών δυνάμεων, ε, για τις περιπολίες συγκεκριμένα, έχει συμμετέχει και η Βρετανία. Διότι μην ξεχνάμε ότι είναι και το πρώτο σημείο επαφής, ε, δηλαδή ε, ενημερώνει την κυβέρνηση για το τι θέλουν οι άνθρωποι όταν είναι θετική η επαφή, δηλαδή όταν δίνεται η εντύπωση ότι υπηρετεί η αστυνομική δύναμη, είναι στην υπηρεσία του, του λαού και όχι, δεν λειτουργεί κατασταλτικά, αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Προσπαθούμε λοιπόν στα πλαίσια των επιχειρήσεων και των μεταρρυθμίσεων των αστυνομικών δυνάμεων να επιτύχουμε και αυτό. Τώρα, ε, στα πλαίσια διαφόρων ε, επιχειρήσεων που έχουμε, ε, η και ζήτημα πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αυτό συνδέεται και με τις αστυνομικές δυνάμεις ε, και χρειάζεται κάποια νομιμοποίηση δεν το σχολήσα νωρίτερα, ίσως έχουμε και στο μέλλον ευκαιρία να το συζητήσουμε. Ε, πρέπει να συνδέσουμε τη μεταρρύθμιση του νομικού ε, συστήματος, του δικαστικού συστήματος ε, με τη μεταρρύθμιση των αστυνομικών δυνάμεων, ε, διότι χρειαζόμαστε την αστυνομία, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, ο εισαγγελέα πρέπει να κάνει ε, τη, δουλειά του, όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά χρειαζόμαστε και οριζόντιες προτάσεις και λύσεις στα πλαίσια μιας σε εντολή θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, παραδείγματος χάρη. Έχουμε το την αντιπροσωπεία η οποία ασχολείται με το θέμα των εισαγγελέων, με το θέμα ε, των ε, υπηρεσιών των πολιτών, δηλαδή με την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία θα συνεργαστούμε στενά ούτως ώστε να ε, προωθήσουμε αυτή την αστυνομική συνιστόση αλλά σας ξαναλέω χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση, οριζόντια προσέγγιση, διότι θα πρέπει όλοι να υπάρχει καθολική υπηρεσία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να δίνουμε την εντύπωση ότι ε, υπηρετούμε ε, πραγματικά τους ανθρώπους ε, και καλύπτουμε τις ανάγκες τους. Η κυρία Φωτήγα, ναι, ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε... Α, η κυρία Νεπόψη, συγγνώμη. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την κατάσταση επιτόπου για την αστυνομία, τις αστυνομικές δυνάμεις. Βεβαίως, θέλουμε περιπολίες να έχουμε σε όλες τις πόλεις. Και γιατί είναι σημαντικό να αρχίσουμε με αυτό, διότι είναι ε, ορατό. Είναι δύσκολε οι μεταρρυθμίσει και οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, λοιπόν, αυτό είναι κάτι απτό. Είναι πρώτο σημείο επαφή. Ε, εάν δουν ε, διαφορετική στάση από πλευρά των αστυνομικών οι άνθρωποι, βοηθάει αυτό πολύ. Για τι εκλογέ βάσει συμφωνία του Μίνσκ και για την κατάσταση στην Ουκρανία. Πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσει μα ε, γιατί μας έχουν απευθυνθεί και κάποιες κατηγορίες. Από πέρσι ε, την οικεχηρία την έχουμε ε, τηρήσει. Εμείς δεν απαντούμε στα πυρά. τα δικά τους, οπότε πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Απόσυρση, ε, αφοπλισμός. Εμείς το κάναμε. Ο, ο, ο ΑΣΕ είπε ότι βρήκε ε, βαρέα πυροβολικά στο Ντονέτσκ, παραδείγματος χάρη. Μην ξεχνάμε, καθημερινά στέλνει νέα όπλα ε, στη δική μας επικράτεια η Ρωσία, οπότε Ε, έχουμε πληροφορίες για 9.500 Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία. Επίσης, 34.000 ε, ε, δυνάμεις των αποσχιστικών δυνάμεων. Τι άλλο να κάνουμε. Μέχρι τα τέλη του 2015 το Κομιτέρνοφ που ήταν στην γκρίζα περιοχή καταλήφθηκε πάλι από Ρώσους στρατιώτες. Υπάρχουν και ε, επιθέσεις. Σύνταγμα. Ναι, δεν θέλουμε να μας κατηγορούν ότι δεν κάνουμε τίποτα, διότι ψηφίσαμε στην πρώτη ανάγνωση κιόλας και το πληρώσαμε με ανθρώπινες ζωές. Παρότι ε, δεν τηρείται πάντοτε η εκεχηρία, θα πρέπει εμείς ε, να δίνουμε το στίγμα μας και ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν τηρούν την εκεχηρία, δεν εφαρμόζεται η συμφωνία, δεν έχουμε ε, αποτελέσματα από ρωσικής πλευράς. Περιμένει η πρόταση για το Σύνταγμα. Θέλουμε να το ψηφίσουμε, αλλά πρέπει να κινηθεί και έλπρεπε να κάνει ένα βήμα προς την πλευρά μας δεν μπορεί να κατηγορεί την Ουκρανία και να ζητάει από εμά μόνο κινήσει για την αμνηστία. Σωστό και δίκαιο το ερώτημα. Να χορηγηθεί. Γίνεται όμως να, να τη χορηγήσουμε σε όλους. Για το MI70 παραδείγματος χαρή Για τις φαγές του Λοβάτ δεν μπορεί να δοθεί συνολικά αμνηστία. Μόνο κατά περίπτωση μπορεί να χορηγηθεί, όχι ε, συνολικά. Για την εφαρμογή, για την αμνηστία για τις τοπικές εκλογές, φυσικά θέλουμε να προχωρήσουμε. Κάναμε τις προτάσεις μας και ακολουθούμε πιστά τη Συμφωνία Μίνσκ. Και όντως θέλουμε να εφαρμοστούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε? Ο Ζαχάρε Κούτσουμ, ο, φυγός της Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, ε, που αναγνωρίζεται μόνο από τη, τη, τη Ρωσία, ενημερώθηκε και ανέφερε ότι θα το λάβει υπόψη Δεν μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε, πρέπει να τους ζητάμε, να ζητάμε από τη Ρωσία να μας αποδείξουν τι κάνουν. Μόνο με συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορούμε να ε, συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σα είπα ότι ψηφίσαμε στην πρώτη ανάγνωση. Έχουμε πρότυπα για να χορηγήσουμε κατά περίπτωση αμνηθία. Έχουμε ε, για, πρόβλεψη για τις τοπικές εκλογές. Αποκέντρωση. Και αυτό το έχουμε. Στην πράξη υπάρχουν αυτά. Περιμένουμε όμως αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά να κάνει κάτι. Για το δεύτερο σημείο, είναι μονόδρομος η Συμφωνία του Μίνσκ. Μονόδρομος αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο της ειρήνης. Και εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να είναι ειρηνική η λύση. Πρέπει να κλιμακώσουμε την πίεση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για άρση των κυρώσεων το καλοκαίρι επειδή υποτίθεται ότι εφαρμόζεται η Συμφωνία του Μίνσκ. Εμείς το ευχόμαστε, το ελπίζουμε και τότε ναι, να έρθουν οι κυρώσεις. Πρέπει να καταλάβουμε τι έχει σημασία εδώ. ασχολούμαστε μόνο με τις κυρώσεις ή μας ενδιαφέρει το μέλλον συμφωνίας ε, του Μίνσκ. Αν ναι, αν μας ενδιαφέρει η συμφωνία του Μίνσκ, περιμένουμε από τα αποτελέσματα από τη Ρωσία. Πρέπει να αποφευθεί η χρήση των όπλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Στέλνουν όπλα Θέλουν στρατιώτες, ένοπλες δυνάμεις. Σε αυτές τις περιοχές ε, πρέπει να είμαστε ετοιμότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, θα το αποφύγουμε. Για να το στείλουμε πολεμοφόδια για, να, για αυτοάμυνα, ποιος δεν θέλει να έχει τη δυνατότητα να ε, αμυνθεί. Και άρα καλό είναι να έχουν πολεμοφόδια. Για τον ΟΑΣΕ στο, στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας βάσει της Συμφωνίας Μίνσκ πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρη την επικράτεια που ακόμη και αυτή που προσωρινά δεν ελέγχει η Ουκρανία. Δεν χορηγείται όμως αυτή η πρόσβαση στη μεθόριο. Ξέρετε ότι τον περασμένο μήνα ε, συζητήθηκε η δυνατότητα να μπορέσει ο ΑΣΕ ε, να ε, έχει πλήρη πρόσβαση για τις μεθοριακές περιοχές ε, απέριφθη από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε μια συμφωνία, ε, σε μια εφαρμογή της συμφωνίας θέλουμε να παίξει αυτό το βασικό ηγετικό ρόλο ο ΑΣΕ, πρέπει να το επιτρέψουμε, λοιπόν. Για την προετοιμασία των τοπικών εκλογών πρέπει να δούμε πώς θα κατοχυρώσουμε την ασφάλεια. Ο ΑΣΕ μπορεί να παρακολουθήσει τις εκλογές μόνο. Αυτή είναι η εντολή του. Ή θα πρέπει να την τροποποιήσουμε την εντολή ή να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα επιχείρησης ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Φυσικά θα αλλάξουν οι εφαρμοστικοί όροι. Ίσως αυτό είναι όμως το επόμενο βήμα που πρέπει να εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ενημερώνουν ότι ήδη είναι παρόν ο επόμενος ομιλητής μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κλείσουμε ε, τούτη τη συζήτηση. Ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που λάβαμε σχετικά με την παρούσα κατάσταση στην Ουκρανία όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, της Συμβουλευτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε σύντομα να μπορούμε πάλι να έχουμε συνάντηση με τον επικεφαλής ε, της αποστολής ε, και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επιχείρηση αυτή. Ευχαριστώ.